Uh, Συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αρχίζουμε παρακαλώ. Καθίστε. I would like to open, um, for those of you who are not from Εγώ είμαι η Ντανούτα Φίμπνερ, για όσου δεν με ξέρουν, που δεν είναι από το Κοινοβούλιο. Είμαι επικεφαλή τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η Σεσίλια Βίξτρομ, που κάθεται δίπλα μου, θα αναλάβει αργότερα, είναι συμπρόεδρος, γιατί είναι πρόεδρος της δεύτερη επιτροπής με την οποία συνεργαστήκαμε για την ακρόαση αυτή. Είναι δηλαδή η δεύτερη επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών. Τώρα δεν θα καλωσορίσω κανέναν, είναι πολύ μακρός ο κατάλογος. Χαιρόμαστε όμως που έχουμε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα θεσμικά όργανα έχουμε και τον Φρανς Τίμερμανς, ε, ε, η πρόεδρο της Επιτροπής. Έχουμε πολλούς διακεκριμένους και έμπειρους ε, προσκεκλημένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη ή μάλλον με λύπη μου σας ενημερώνω ότι επειδή ήταν, είναι υψηλό το επίπεδο ασφάλειας, έχει τώρα αναβαθμιστεί στο Κοινοβούλιο το επίπεδο συναγερμού και ασφαλείας, είχαμε προβλήματα στις προσκλήσεις και πολλοί δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να έρθουν όλοι όσοι ήθελαν να έρθουν στην ακρόαση αυτή και να παρευρεθούν. Όμως ε, αναμεταδίδεται η συνεδρίαση, υπάρχει web streaming και έτσι στο διαδίκτυο μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να ε, παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Μπορούν. Και υπάρχει και hashtag για αυτή την ακρόαση. Ίσως να το έχετε και εσείς ήδη λάβει. Είναι hash, EP, hearing, on, ECI, hash. Θα ήθελα για λίγα λεπτά να σας εξηγήσω ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα θεωρούσαμε ότι το ΠΕΠ, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, είναι πολύ άμεση και πρακτική έκφραση ε, της νέας διάκρισης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης. Ως θεσμικά όργανα εμείς τώρα είμαστε στη διαδικασία ε, ε, ενσωμάτωσης αυτής αυτών των νέων ε, δεδομένων με βάση τα οποία μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν και να είναι μέρος της διαδικασίας λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων. Έτσι προετοιμαζόμεθα καλύτερα για να αντιδρούμε και να επεξεργαζόμεθα τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών ανδρών και γυναικών. Οι περισσότερες προσδοκίες εκφράζονται μέσα από την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωή και έχουν πολλέ διαστάσει, όπω αηφορία, διατηρησιμότητα στην Ευρώπη μετά την κρίση. Εμεί ω Κοινοβούλιο στηρίζαμε την ΠΕΠ ω στοιχείο κλειδί που εξοπλίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Μια ευκαιρία οι Ευρωπαίοι πολίτες να γίνουν μια συνιστόσα εξουσία, όχι μια εξουσία που μόνο επικυρώνει τις αποφάσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω και κάτι που δεν το ακούμε συχνά, ούτε το λέμε συχνά, αλλά χάρη στην ΠΕΠ, την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, βλέπουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι αλήθεια ότι αδιαφορεί ο κόσμο για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για το πώ διαμορφώνεται η Ευρώπη. Γιατί και η Σεσίλια Βίξτρομ και ο Φραν Τίμερμαν θα μα τα πούν αυτά, αλλά αν κατάλαβα καλά, 49 πρωτοβουλίε ε, άρχισαν, δηλαδή περίπου 8 με 10% του πληθυσμού της Ευρώπης συμμετέχει. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που δεν είναι αδιάφοροι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουν ε, δραστήρια να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν την Ευρώπη. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν για ποιο σκοπό υπάρχει η Ευρώπη και τα θεσμικά της όργανα. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Ε, εμείς ε, βλέπουμε ε, να υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες και η συμμετοχική δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι διαφορετικές αυτές προσδοκίες όπως προέρχονται από τα διαφορετικά σημεία της Ευρώπης. Έτσι εκφράζεται το τι περιμένει ο κόσμος από την Ευρώπη. Τώρα, η Σεσίλια θα συνεχίσει, αλλά έχω και τον Κάρλο Καζίνη εδώ. Δεν ξέρω, κάνω μια εξαίρεση, δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό. Θέλω να καλωσορίσω κάποιον που είναι πολύ σημαντικός για μας και που εργάστηκε και οικοδόμησε επί χρόνια την Επιτροπή, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής μας. Καλώς ήρθατε κυρία Καζίνη, χαιρόμαστε που μπορέσατε να έρθετε. Και τώρα Σεσίλια έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ντανούτα. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να σας καλωσορίσω όλους τους φίλους, τους συναδέλφους, τους ομιλητές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την ακρόαση για την ε, υλοποίηση του και την εφαρμογή του κανονισμού πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών, μια ακρόαση που συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και Αναφορών. Όπως ξέρετε, η, Ευρωπαϊκή, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών υπάρχει από την 1η Απριλίου του 2012 όταν ο κανονισμός ε, ε, τέθηκε σε ισχύ. Ο σχετικός κανονισμός. Με αυτόν τον κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα εργαλείο ένα μέσο που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε στην ε, διαμόρφωση του κανονισμού ΠΕΠ από την ευθύνη εξ αρχής ως σχετική επιτροπή συνεργαζόμενη στενά με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα καλής συνεργασίας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2010... Η Νταϊάννα Wallis που ήταν η εισηγήτρια στην Επιτροπή Αναφορών και χαίρομαι που την καλωσορίζω και κάνω και μια εξαίρεση στα καλωσορίσματα και εγώ, είναι θαυμάσιο που βρίσκεσαι εδώ. Μαζί με την ε, Γκέραντα Χόφνερ ε, συνεργάστηκαν και τον Αλέν Λαμασούρ και την ε, Ζήτα Γκουρμάη που ήταν εισηγητές από την Επιτροπή ΑΦΚΟ, συνταγματικών υποθέσεων. Καλώς ήρθατε όλοι και συνεργάστηκαν για να γίνει φιλικό προς τους πολίτες το μέσον αυτό αλλά και να είναι και αποτελεσματικό. Ο κύριος Μπεσέρα είναι ο συντάκτης από την Επιτροπή ΠΕΤΗ και ήδη άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα για να βελτιωθεί το σχετικό μέσο καλύτερα μαζί με την ε, κυρία Σέπφλιν από την Επιτροπή ΑΦΚΟ ε, που είναι η συγκήτρια. Καλή συνεργασία και καλή επιτυχία. Τώρα πρέπει να, με τρία χρόνια μετά να δούμε προσεκτικά το πώς εφαρμόστηκε αυτό το διάστημα ο κανονισμός. Είπαμε, 50 πρωτοβουλίες υπευλήθησαν στην Κομισιόν, η ΠΕΠ έδειξε ότι έχει μεγάλη δυναμική και πολλές δυνατότητες, ε, αλλά φαίνεται ότι τώρα ε, μειώνεται λίγο αρχικός ενθουσιασμός και ε, δεδομένων κάποιων βασικών προβλημάτων. Η κριτική αφορά την έλλειψη διαφήμισης και σαφή ενημέρωση σχετικά με το ΠΕΠ, την έλλειψη πόρων, και τους επαχθείς όρους ε, που αφορούν τις δηλώσεις υποστήριξης. Όλα αυτά είναι εμπόδια τα οποία ε, παρενοχλούν και μειώνουν τη συμμετοχή των πολιτών. Καθήκον μας είναι λοιπόν να βρούμε τα καταλληλότερα και αποτελεσματικότερα μέσα για να βελτιώσουμε αυτή τη δυνατότητα που δίνει μια ισχυρή φωνή στους πολίτες. Αυτό χρειάζεται αυτούς τους καιρούς στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Αναφορών έχει ε, διεξοδική και μεγάλη πείρα ε, από τους πολίτες και την επαφή με εκείνους. Ε, τους προσκαλούμε, τους δίνουμε το λόγο και η φωνή τους έτσι φτάνει του υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, συγκινητικό και αποτελεσματικό. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Ε, Επίση, εξετάζονται οι πρωτοβουλίε που δεν μπορούν να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό, γιατί δεν έχουν ακολουθηθεί όλε οι σχετικέ και απαραίτητε διαδικασίε. Θα ακούσουμε σήμερα την εμπειρία των οργανωτών από τις λεγόμενες αποτυχήσεις ε, πρωτοβουλίες. Μία από αυτές είναι το ECOSIDE, η οικολογική καταστροφή. Υποθέτω ότι οι δύο επιτροπές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον, Ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θα εξετάσουν τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να συνεχίσουμε αυτό το τόσο πολύτιμο δημοκρατικό μέσο. Τώρα έχω τη χαρά και την τιμή να δώσω το λόγο στον Φρανς Τίμερμαν, πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να έχετε υπόψη σας ότι ο κύριος Τίμερμαν είναι, είναι ο επιτροπός μας στην Επιτροπή Αναφορών. Για πρώτη φορά έχουμε επίτροπο και είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να σας καλωσορίσουμε στην ακρόαση αυτή. Να θυμίσω επίσης στους συναδέλφους ότι ο Επίτροπος Τίμερμανς θα παρευρεθεί στις 15 Μαΐου στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΕΤΗ το απόγευμα. Και θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε διάλογο και να μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε για αυτά. Σήμερα ο κύριος Στίμερμανς ήρθε εδώ για να ακούσει τη, κυρίως την εμπειρία των οργανωτών και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα το λόγο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ως επίτροπός σας... Είμαι επίτροπος όλων κυρίε και κύριοι. Ή τουλάχιστον θα ήθελα να είμαι. Βλέπω μάλιστα πρόσωπα που τα βλέπω εδώ και 10 χρόνια. Όταν για πρώτη φορά αρχίσαμε να μιλούμε για πρωτοβουλίες των πολιτών και υπήρξε μεγάλη αντίσταση σε αρκετά κρατημέλη σχετικά με αυτό. Επιμείναμε, εργαστήκαμε, αρκετοί από εσάς το ξέρετε αυτό, ξέρετε τι προσπάθεια καταβάλαμε. Και συμφωνώ με τις επικρίσεις, δεν έχουν γίνει όλα τέλεια, αλλά και εγώ θεωρώ ως πρώην υπεύθυνο ότι πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα. Πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία που οδηγεί στις πρωτοβουλίες των πολιτών ώστε να παραμένει στις προθέσεις των ανθρώπων και να δημιουργεί μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Αυτό το λέω κατανοώντας απολύτως ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μια τεράστια απόκληση μεταξύ του τι συμβαίνει σε θεσμικό πλαίσιο και του πώς γίνεται αυτό αντιληπτό στην κοινωνία την ευρωπαϊκή. Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης στις κοινωνίες μας, στις χώρες μας, μεταξύ ομάδων εθνικών, ενώσεων, γενεών και αυτό προβάλλεται πιο μακριά και ευρύτερα όταν βλέπει κανείς το ευρωπαϊκό επίπεδο, το θεσμικό. Και βεβαίω μια πρωτοβουλία των πολιτών δεν μπορεί να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Θα ήταν ανόητο να πιστεύει κανείς ότι μια πρωτοβουλία μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τόσο ευρύ και τόσο σοβαρό που αφορά σε όλες μας τις κοινωνίες. Τώρα βέβαια είναι μία, ένα από τα λιθαράκια που θα οικοδομήσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη. Η Κομισιόν θα υποβάλει μια έκθεση για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών μέχρι τον Απρίλιο. Και εγώ θα ήθελα να σας ακούσω σήμερα πολύ πολύ προσεκτικά. Δεν θα είναι δυνατόν να είμαι συνεχώς παρόν σε όλη την ακρόαση γιατί έχω πολύ φορτωμένη μέρα σήμερα αλλά σας υπόσχομαι ότι τα σχόλιά σας θα διαβιβαστούν από τους συναδέλφους και θα ενσωματωθούν στην έκθεση που θα υποβληθεί μέχρι τον Απριλίο. Και η προσωπική μου δέσμευση είναι ότι θα αναζητήσω νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που ανέφερα πριν την έλλειψη εμπιστοσύνη, την έλλειψη ενθουσιασμού και για πολιτικούς και για πρακτικούς λόγους. Και όπως έλεγα εδώ στο Κοινοβούλιο, στην αρχή τη θητείας μου, στην ακροματική διαδικασία, εγώ θα ήθελα να ακολουθήσω μια πολιτική προσέγγιση και οδό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν νομικοί λόγοι γιατί η Κομισιόν θα μπορούσε να λέει ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία που δεν μπορεί να υποβληθεί και τα αλλά αυτό δεν πρέπει να αποθαρρύνει. Γιατί ακόμα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοια πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα διαλόγου και να συνεχιστεί ο διάλογος αυτός. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε προσεκτικά τον κανονισμό, θα πρέπει να εκτιμήσουμε κατά πόσον πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί στην πραγματικότητα τα μόνα όρια που τίθενται είναι τα όρια που θέτει η συνθήκη. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την όποια ευελιξία έχουμε ώστε να δώσουμε μια μεγαλύτερη πολιτική όθηση σε αυτό το πολύ σημαντικό μέσο διαλόγου με τους ε, πολίτες της Ευρώπης. Και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διευρύνουμε τη γνώση σχετικά με την πρωτοβουλία, την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον στην κοινωνία. Θα πρέπει να είναι γνωστή από περισσότερους πολίτες στην Ευρώπη. Και απλώς κλείνω λέγοντας ότι είμαι εδώ για να σας ακούσω, για να βελτιώσω το μέσο όσο γίνεται εντός των ορίων και των δυνατοτήτων της συνθήκης. Συνεχίστε, σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε το διάλογο και ίσως και η έκθεση που θα υποβάλουμε τον Απρίλιο να είναι το επόμενο βήμα για την οικοδόμηση αυτού του διαλόγου. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, Αντιπρόεδρο και θα πάμε τώρα στους ειδικού εν πάση περιπτώσει. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Θεντέγιας που είναι εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας Right to Water που είναι μία από τις πρώτες επιτυχείς πρωτοβουλίες. Ε, θα ήθελα να ζητήσω τα δικά σας σχόλια. Τώρα ξέχασα το πιο σημαντικό. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Ας προσπαθήσουμε όλοι με να είμαστε σύντομοι για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ο κύριος Τεντέγιας. Ναι. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. να παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία Right to Water. Εγώ είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της πρώτης επιτυχούς τέτοιας πρωτοβουλίας. 1,9 εκατομμύρια υπογραφές συλλέξαμε με ψηλό ποσοστό επικύρωσης και ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε συλλέξει 1 εκατομμύριο από 7 χώρες μέχρι τα μέσα του 2013. Υπάρχει λοιπόν μια νομιμοποίηση, μια κάποια νομιμοποίηση για να μιλήσουμε για προβλήματα, προκλήσεις, λύσεις που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβουλίες και συμφωνώ με τον κύριο Τίμερμανς ότι είναι κυρίως πολιτικό θέμα πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες που είμαι βέβαιος ότι με καλή θέληση μπορούμε να υπερβούμε. Εμείς αναφερόμασταν στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό με όλες του τις χρήσεις και με τις χρήσεις για την υγιεινή, έτσι όπως είχε οριστεί από το 2010, το να εξαιρεθεί αυτό από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και από εμπορικές συμφωνίες κυρίως, και να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στο νερό καθιδρύοντας αυτό το δικαίωμα, το ανθρώπινο δικαίωμα στο είδωρο καθώς προχωρούμε και με τους στόχους της χιλιετίας. Πρόκειται πράγματι, όπως είπατε και εσείς, για ένα θέμα εμπιστοσύνης και έχοντας ασχοληθεί ένα χρόνο τώρα έχουμε λάβει ανταπόκριση από την Κομισιόν, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες κτλ. Μας λείπει ακόμα μια δεσμευτική νομοθεσία που θα μετέτρεπε το αίτημά μας σε δεσμευτική διάταξη. Νομίζω ότι εμπίπτουμε στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης. Βεβαίως όπως είπατε και εσείς ε, δεν είναι τέλειο το εργαλείο αυτό, το μέσο αυτό. Αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα διακρατικό μέσο, δημοκρατικό, δεν είχαμε και πολλά σημεία αναφοράς και σύγκρισης, Είμαι βέβαιος ότι μπορούν να επιληθούν τα τεχνικά και νομικά προβλήματα, αλλά είναι ένα ορισμονισμένο πρόβλημα συλλογής υπογραφών, για παράδειγμα, online, θα βοηθούσε. Αλλά βέβαιως ε, χαιρετίζω και το έργο της Κομισιόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να βελτιωθούν αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Όπως έλεγα όμως ε, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη δεσμευτικών διατάξεων κάτι δηλαδή απτό το οποίο να μας έδινε η Κομισιόν που να έθετε ένα πλαίσιο. Υπάρχει η έκθεση που αναφερθήκατε και εσείς για το νομικό πλαίσιο των ε, πρωτοβουλειών πολιτών και έχουμε και επί του περιεχομένου της πρωτοβουλίας ε, συζητήσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο, όπως και στο παρελθόν, θα είναι σύμμαχος. Σύμμαχός μας για να προωθήσουμε τις, ε, τα αιτήματα σχεδόν 2 εκατομμυρίων πολιτών που έχουν υπογράψει. Υπάρχει προφανώς ενδιαφέρον από πλευρά των πολιτών για τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές, τις ενωσιακές πολιτικές. Αλλά εάν αυτή η συμμετοχή είναι μόνο συμβουλευτική και μόνο όταν σας αρέσει και σας βολεύει, τότε το χάσμα μεταξύ θεσμών και πολιτών θα αυξηθεί, θα μεγαλώσει. Και επομένως το μέσο των ECI, των Πρωτοβουλίων των πολιτών, είναι ένα μέσο το οποίο αντιμετωπίζει κάποιους περιορισμούς ε, αυτή τη στιγμή, αλλά είναι στο χέρι μας της Κομισιόν του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι αυτοί οι λίγοι χαρακτήρες που μας επιτράπει να τοποθετήσουμε στο κείμενο πρέπει να αντιμετωπιστούν από εσάς ως, ως πολύτιμος λήθος για να βοηθήσουμε τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη 20 δευτερόλεπτα εγκλίνω ε, ε, ε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια τα τελευταία λίγα χρόνια έχει εστιαστεί σε θέματα καλύτερης ε, νομοθεσίας ενώ θεωρούμε ότι θα έπρεπε να εστιαστεί στην καλύτερη δημοκρατία, το οποίο δεν είναι ένα αγαθό που έρχεται με υψηλό κόστος, είναι ένα απόλυτο πλεονέκτημα και θα πρέπει λοιπόν να υποστηριχθούν καλύτερα, περισσότερο οι διοργανωτές τέτοιων πρωτοβουλειών ώστε το μέσο να είναι πιο user-friendly όπως λέμε στα ελληνικά. Επομένως, από την Κομισιόν εξαρτάται να διακηρύξει ότι το είδωρ είναι ανθρώπινο δικαίωμα και να μην το αποκλεί αυτό το γεγονός από εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτική της ανάπτυξης να συμπεριλαμβάνει και την πτυχή και το επίπεδο του νερού. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, ευχαριστώ να ήμουν αρκετά σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Σεμπέλιος. Ε, δεν είναι ίσως ε, παρηγοριά, αλλά ε, θα έχετε και αργότερα δικαίωμα να μιλήσετε, μιλήσατε αρκετά και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Πρίσκα Μέρτς. Εσείς διευθύνετε την Ecoside in Europe που είναι πρωτοβουλίες που έχουν αποτύχει και να δούμε ποιος είναι ο δρόμος προς την επιτυχία να μας πείτε γιατί, ε, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία για ορισμένες ε, πρωτοβουλίες. Ε, θα μπορούσα να έχω τις διαφάνειες ίσως. Τις έστειλα. Τις έστειλα παντού. Κρίμα. you go Να αναφερθείτε βέβαια στην παρουσίαση. Αρχίζω, κύριε ε, Επίτροπε, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, διότι νομίζω ότι ήταν απαραίτητη. Νομίζω ότι το 2012 ήμασταν μια μικρή ομάδα ατόμων και η ε, ιδέα του EcoSide ε, μας ενδιέφερε και πιστεύουμε στην δημοκρατία στην Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι δύσκολο να μαζέψει κανείς ένα εκατομμύριο υπογραφές. Μήπως μιλάω γρήγορα. Ε, δύο χρόνια αργότερα ξέραμε ότι είχαμε, ε, είχαμε σφάλει και ότι το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο ε, και η δημοκρατία στην Ευρώπη δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Πρέπει όμως να έχει ακόμα τις δυνατότητες να, <clears throat> να μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δημοκρατία. Ε, το πρώτο αρνητικό σημείο είναι ότι πάρα πολλοί πολίτες αποκλείονται από συμμετοχή σε πρωτοβουλία. Αυτοί που ζουν στην Πορτογαλία, στην Αυστρία δεν μπορούν <clears throat> και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχουν ένα δικαίωμα και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να το ασκήσουν. Όσοι ε, έχουν, δεν έχουμε ε, πρόσβαση στι στατιστικές. Το ιστότοπός μας ε, στις στατιστικές του μας δείχνει ότι μόνο 44% αυτοί που κλικάρουν χάδονται στην διαδικασία και δεν μπορούν να υπογράψουν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι προϋποθέσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία έχουν δυσκολίες. Πώς λοιπόν μπορούμε να κρατήσουμε τα κίνητρα στην ομάδα μας όταν δεν έχουμε αποτελέσματα και έχουμε απάντηση από την Κομισιόν που μας λέει ότι η διαδικασία γίνεται ευκολότερη, αλλά δεν γίνεται ευκολότερη, αντίθετα γίνεται χειρότερη. Θα πρέπει η διαδικασία να είναι φιλική προς τους πολίτες, προς τα άτομα με αναπηρίες για να μπορούν να υπογράψουν. Ε, θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικές ε, υπογραφές, ε, να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο προσβάσιμο. Και ακόμα και η πιστοποίηση του συστήματος συλλογής είναι πάρα πολύ δυσχερής και είναι περίπου αδύνατον αν δεν έχει κανείς τις νομικές γνώσεις να ακολουθήσει την διαδικασία το έντυπο διότι αν πηγαίνει κανείς σε μια εκδήλωση διεθνή και πρέπει να πάρει 28 διαφορετικά έντυπα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε, έχουμε μια ταυτότητα ευρωπαϊκή, θα πρέπει να έχουμε ένα έντυπο για να υπογράψει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Το θέμα του χρόνου επίσης είναι σημαντικό είναι ένα πρόβλημα πρακτικό. Δεν υπάρχει χρόνος ανάμεσα στην ε, εγγραφή ε, και είναι δύσκολο να προγραμματίσει κανείς, να οργανώσει προβολή στα μέσα ενημέρωσης, να οργανώσει το θέμα για την πρωτοβουλία. Πρέπει να υπάρχει μια περίοδος έξι μηνών μετά την καταχώρηση για να μπορεί κανείς να προετοιμάσει την όλη πρωτοβουλία. Επίσης μας ανησυχεί το γεγονός και βλέπετε εδώ ότι ε, τι ε, λύπη βλέπουμε στο τέλος. Οι υπογραφές είναι αρκετά σημαντικές. Αν είχαμε λοιπόν περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να οργανώσουμε καλύτερα την πρωτοβουλία. Μας ανησυχεί το ε, ε, το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μια νομική προσωπικότητα ή ίσως ΜΚΟ ευρωπαϊκές για να περιορίσουμε ε, την ευθύνη, την ευθύνη των ατόμων. Αν πρέπει κανείς σε 28 χώρες να είναι υπεύθυνος, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο Έχουμε μεταφράσει τη μεθοδό μας σε πάρα πολλές γλώσσες ευρωπαϊκές. Έχουμε διαδώσει όλο το κίνημα ε, διασυνοριακά και τώρα εξακολουθούμε να είμαστε Ευρωπαίοι και διεθνείς. Μπορεί λοιπόν τη ε, πρωτοβουλία να είναι πάρα πολύ χρήσιμες και έχουμε 12 βήματα που προτείνουμε ούτω ώστε να επιτύχει κανείς με την πρωτοβουλία σχετικά με το μέλος. Ε, έχουμε πάρα πολλά εκατομμύρια πολιτών, αλλά πάρα πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι διότι έχουμε ανεργία, έχουμε συρρήκνωση του κράτους, έχουμε υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο θέμα των τραπεζών. Ε, Πάρα πολλοί λοιπόν δεν ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα ψήφου στις εκλογές. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία των πολιτών των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, να δεχθούμε, να χαιρετήσουμε το διάλογο για τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για μας τους πολίτες. Και υπό το φως αυτών οι τάσεις απόρριψης ορισμένων επίμαχων πρωτοβουλειών είναι κάτι το ανισχυτικό. Γιατί πρέπει ο έλεγχος να γίνεται στην αρχή. Και έχω, πρέπει να έχουμε μια ατζέντα, να μπορούμε να επιλέξουμε η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Ε, διέρχεται μια μεγάλη κρίση. Ας μην στερήσουμε αυτούς ε, που ζουν στην Ευρώπη να χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Τότε εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορούν να απευθυνθούν στους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς και θα ε, αναθερμανθεί ήδη ο δημόσιος διάλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες και θα έχουμε μια, ένα νέο νόημα για το εγχείρημα ειρήνης ε, στην Ευρώπη. Είναι στα χέρια σας να οικοδομήσουμε αυτό το σύστημα πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών που να λειτουργεί καλά και να έχει επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Θα θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να περιορίζετε στα πέντε λεπτά, διότι δυστυχώς ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ο κύριος Γιώχανσον είναι ε, δικηγόρος και εκπροσωπεί το Minority Safe Pack Case. Im Juli 2013 haben die in το 2013 οι οργανωτές για την πρωτοβουλία αυτή μάζεψαν τις, ε, το 1 εκατομμύριο υπογραφές για την προστασία των μειονοτήτων στην Ευρώπη. Οπότε τέθη το αίτημα καταχώρησης ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή δύο μήνες αργότερα απερίφθη η πρόταση με τη δικαιολογία ότι βρίσκεται εκτός του πλαισίου μέσα στο οποίο είναι εξουσιοδοτημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη. Η απόρριψη δεν ήταν ούτε δύο σελίδες. Το 2013 εγώ προσέφυγα στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου για έφεση και κατέθεσα την έφεση στα γερμανικά. Τρία κράτη-μέλη κατόπιν έθεσαν έτοιμα ούτω ώστε ε, να συμμετέχουν στη διαδικασία. Η Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρουμανία ε, είναι οι χώρες ε, από τις οποίες προέρχονται ή παρεμβαίνονται στο δικαστήριο. Η Ρουμανία απεσύρθη απεσηρθη αλλα ε, διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στην προφορική διαδικασία. Η υπόθεση στις 25 Νοεμβρίου του 2013 ε, εκδικάστηκε ε, ε, ε, κατεχωρήθη στο δικαστήριο. Με την πρωτοβουλία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των γλωσσικών μειονοτήτων, να βελτιώσει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν και να ενισχύσει την πολιτιστική διαφορετικότητα προβαίνοντας στην θέσπιση νομικών πράξεων για τη βελτίωση όλων αυτών. Ε, και διασφαλίζοντας ή ενισχύοντας την ε, διαφορετικότητα. Αυτά τα μέτρα αφορούν τις μειονότητες, τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους, τη συμμετοχή τους, την ισότητα, οπτικοακουστικά μέσα ε, στην υπηρεσία τους, άλλα μέσα από τα ΜΜΕ ε, και μέτρα πρόθεσης από το κράτος. Η καταχώρηση απερίφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να γίνει πρόθεση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό είναι πολύ αξιοπερίεργο. Ο κανονισμός μας είπαν ότι προβλέπει, προβλέπει όμως ότι όλες οι ε, καμία ε, πρόταση δεν θα καταχωριστούν. Ε, επίσης θα πρέπει αναφέρθηκε ότι δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι όμως ανεπαρκής η αιτιολόγηση. Υπάρχει η ένσταση ότι παραβιάζεται το άρθρο 296 και το άρθρο 4 ε, των σχετικών κανονισμών. Οι ε, ε τούντες αναφέρουν ότι ε, δεν βρίσκονται εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους και ότι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικές προτάσεις. Είναι, προβλέπεται αυτό με βάση το άρθρο 296. Επίσης προστίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρει γιατί ο κανονισμός 211 του 11 δεν μπορεί ε, να καταχωρήσει μια πρωτοβουλία των πολιτών ή μέρος αυτής. Οι πρωτοβουλίε ε, είναι για τους ε, συνήθεις, τους απλούς πολίτες, όχι για τους νομικούς. Θα πρέπει να μπορεί ο πολίτης να καταλαβαίνει γιατί απορρίπτεται μια πρωτοβουλία του ε, και να μην αντιμετωπίζει μόνο την νομική γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει. Πιστεύουμε ότι η ε, πρέπει να ξαναδούμε ε, το ζήτημα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα και αν ένα από τα θέματα είναι εκτός ε, αρμοδιότητας, μπορεί να περιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρωτοβουλία στα υπόλοιπα θέματα και να, τα να καταχωρήσει την πρωτοβουλία. Ε, όταν μια πρόταση θεωρείται μη παραδεκτή, αυτό δεν μπορεί να έχει επίπτωση στις υπόλοιπες προτάσεις. Στην ε, περαιτέρω διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δώσει μια αιτιολόγηση ε, για την στάση της παραδέχεται όμως για ορισμένες προτάσεις ότι έχει την αρμοδιότητα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα σας δίνω το λόγο. Ας αρχίσω από το τελευταίο αυτό. Αυτό που έκανε ο κύριος Γιώχανσον είναι να παρουσιάσει ε, την ε, ε, θέση του όπως γίνεται στο δικαστήριο. Δεν μπορώ βεβαίως εγώ να ε, κάνω νομικές παρατηρήσεις. Η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο και εκεί ε, θα εκδικαστεί η υπόθεση. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε. Όμως σας άκουσα πολύ προσεκτικά και ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξαναδούμε πάλι το ζήτημα αυτό. Πάντως γενικά Αυτό που θα πλούστευε τα πράγματα στο μέλλον είναι το εξής. Όταν αναλαμβάνετε μία πρωτοβουλία, να εξετάζετε καταρχήν αν η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων, ούτως ώστε να υπάρχει και η αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει επιτυχία σε μία χώρα, παρόλο που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους ε, ε, επιχειρείται να περάσει ε, μέσα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όμως πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει εκεί όπου έχουν αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη, ενώ εμείς όχι. Προσοχή λοιπόν να υπάρχει η διευκρίνηση, η απαραίτητη που θα μας αποτρέπει από παρανοήσεις. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα σημεία στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και στην έκθεσή μας τον Απρίλιο εκεί θα επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Το ίδιο θα ήθελα να πω και σε εσά, κυρία Μέρθ, γιατί πολλά από αυτά που είπατε ε, είναι εύλογα, θεωρώ. Ποτέ δεν ήταν βέβαια πρόθεσή μας να δυσκολέψουμε τους πολίτες από το να συμμετέχουν. Όμως, σε τελευταία ανάλυση, όσα κάνουμε πρέπει να είναι ένομα, να έχουν νομική βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια του νόμου περισσότερο από κάθε άλλο θεσμικό όργανο. Αλλιώς ε, θα γίνει προσφυγή στο δικαστήριο και θα υποστούμε συνέπειες. Κατανοώ λοιπόν την παρατήρηση για την ευελιξία, αλλά υπάρχει κάποιο όριο στην ευελιξία που μπορώ να σας δώσω. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις πολυάριθμες παρατηρήσεις σας και θα φροντίσουμε ώστε η αντίδρασή μας στην έκθεση του Απριλίου να καλύπτει τα θέματα που θέσατε. Μάλλον δεν θα μπορέσουμε να σας καλύψουμε σε όλα τα θέματα που θέσατε, αλλά θα κάνουμε προσπάθειες να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτό είναι το σημείο εκκινήσεώς μας. Τώρα για το νερό. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια επιτυχέστατη πρωτοβουλία. Μέχρι τώρα είναι υποδειγματική για το πώς μπορούμε να δουλέψουμε θετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε πολύ συγκεκριμένα υποβάλλοντας προτάσεις στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας για τη βελτίωση της κατάστασης με έναν αριθμό συγκεκριμένων ε, αποτελεσμάτων. Βέβαια όλα αυτά οριοθετούνται από ε, ε, το σημείο όπου σταματά η εθνική αρμοδιότητα και αρχίζει η ευρωπαϊκή. Ορισμένα θέματα σε σχέση με την πρόσβαση στο νερό δεν ε, είναι αντικείμενο ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά παραμένουν στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας οπότε εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όμως εμείς προσπαθήσαμε να καταπιαστούμε με έναν αριθμό θεμάτων που ε, ετέθησαν στην πρωτοβουλία των πολιτών και αλλάξαμε και ορισμένα στοιχεία στην πολιτική μας για τα ύδατα. Θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση σχετικά με το κράτος δικαίου. Που τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μεταξύ άλλων στο πώς θα παραμείνουμε εντός του νομικού πλαισίου που έχουμε, που είναι δεδομένο. Παράλληλα, το κράτος δικαίου μας δίνει δυνατότητα να δούμε πώς εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη, από τα κράτη-μέλη, ε, με βάση τις εθνικές αρμοδιότητες. Εδώ αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο θέμα των μειονοτήτων. Δεν συμφωνώ με τη δήλωση ότι αρνηθήκαμε να κάνουμε οτιδήποτε για τις μειονότητες. Πολύ συγκεκριμένα Τις τελευταίες βδομάδες ένα από τα θέματα που με απασχόλησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας που αυξάνονται σε πολλά από τα κράτη-μέλη μας. Και παρόλο που δεν είναι όλα ευρωπαϊκές αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε θετικά αρχίζοντας από το ποια είναι η δυνατότητα που έχουμε για να παρέμβουμε στα ζητήματα αυτά. Και θα γίνει ε, μια πρώτη συνάντηση τέλος Οκτωβρίου για τα θέματα αυτά. Το θέμα του θα είναι καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας και την ανάγκη για ανεκτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να δείξουμε ότι οι μειονότητες και τα δικαιώματά τους αποτελούν μεγάλο κομμάτι της βασικής εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορείτε να βασιστείτε σε μένα να προωθήσω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και έχουμε ε, τον κύριο Ιαν Χάρντεν, Γενικό Γραμματέα αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ε, τις απόψεις του διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας ε, τις δύο επίτροπες και την κυρία Χιούμπνερ και Βίλξτρομ που κάλεσαν τον Ομπούτσμαν να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση και δημόσια κρόαση. Η άμεση αντίδρασή μου όταν εξέτασα το πρόγραμμα ήταν πολύ καλά. Έχουμε να κάνουμε με την νομική άποψη, τεχνική και οργανωτική. Τι γίνεται με την πολιτική άποψη του θέματος. Η πραγματική σημασία ε, της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι πολιτική. Εξέτασα τις λεπτομέρειες και είδα ότι πολλοί ευρωβουλευτές θα λάβουν το λόγο και συναντιόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που είναι το πολιτικός θεσμός άμεσα εκλεγμένος από τους πολίτες. Σκεφτόμαστε την δημοκρατία σε δράση που βλέπουμε εδώ σε αυτό το κτίριο σήμερα. Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών είναι μεταξύ των δημοκρατικών αρχών και η λειτουργία της Ένωσης πρέπει να βασίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και οι πολίτες αντιπροσωπεύονται άμεσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία περιγράφεται ως ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας και περιλαμβάνει την συμμετοχή των πολιτών ε, στην δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Και όμως θα ήταν λάθος ε, να ασχολούμαστε μόνο με την αντιπροσωπευτική και συμμετοχική δημοκρατία. Θα πρέπει να ενισχύονται, να αλληλοενισχύονται αμοιβαία στην πρακτική. Η επιτυχία εξαρτάται όχι μόνο από την Επιτροπή αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα επανέλθω στο σημείο στο τέλος της παρουσίασής μου. Το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να υποβάλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θεωρηθεί ως μέσο σημαντικό συμμετοχής των πολιτών μαζί με την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και αν οι πλήρες δυνατότητες του συστήματος της πρωτοβουλίας πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν πλήρως, αυτό ισχύει και για τις αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η αποστολή του διαμεσολαβητή όπως ανακοινώθηκε στην περσινή στρατηγική είναι να ε, συνεργάζεται με τους θεσμούς της Ένωσης για καλή ε, δημοκρατία, για μια διοίκηση ηθική και που θα λογοδοτεί. Ο Ombudsman τονίζει την ανάγκη για την πρωτοβουλία να γίνει ένα μέσο όσο το δυνατόν διαφανές και φιλικό προς τους πολίτες. Στο τελευταίο έτος ε, προσπάθειες έχουν ε, καταβληθεί ε, με αρχικές έρευνες και διερευνητικές εργασίες και η κυρία Τίνα Νίλσον που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό κάθεται εδώ στα αριστερά μου. Στην έρευνα αυτή θέλουμε ο κανονισμός να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός ε, και να έχουμε ε, τροφή ε, και συνεισφορά για το νομοθετικό σώμα στην εργασία που γίνεται φέτος. Προσπαθήσαμε να ρωτήσουμε τις οργανώσεις ποια ήταν η θέση τους να αναλύσουμε τις απαντήσεις τους και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να απαντήσει σε ορισμένα σημεία κλειδιά που θα έχουν καθοριστεί. Ε, να δοθούν αιτιολογήσει εάν δεν θεωρείται παραδεκτή μια πρωτοβουλία. Αν έχει υπάρξει ένα δικαίωμα αμφισβήτησης, αντίθεσης ε, στην πρωτοβουλία. Όσον αφορά το 1 εκατομμύριο υπογραφές, τονίσαμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει σαφώς να εξηγήσει τη θέση της για το θέμα, ακόμα και για την πολιτική άποψη του θέματος. Η σαφήνεια για τα επιχειρήματα των επιλογών προωθούν επικοδομητική συζήτηση ε, την δημοκρατία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήσαμε διευκρινήσεις από την Κομισιόν για ορισμένα νομικά και πρακτικά θέματα. Η απάντηση της Κομισιόν που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και πλήρης υπάρχει στον ιστότοπο του διαμεσολαβητή, της διαμεσολαβήτριας. Ε, θα δημοσιεύσουμε ε, την θέση σχετικά με αυτήν την προκαταρκτική έρευνα τον επόμενο μήνα. Αλλά μπορούμε να συμμεριστούμε σήμερα ε, τις βασικές, ε, τα βασικά πορίσματα. Η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού με φιλικό τρόπο προς τον χρήστη, αλλά η Κομισιόν μπορεί να δράσει μόνο μέσα στα πλαίσια τα νομικά του κανονισμού και είναι λυπηρό, όπως ήδη εξηγήθηκε σήμερα, ότι ε, μερικές διατάξεις του κανονισμού θέτουν εμπόδια ε, νομικά και γραφειοκρατικά ε, σε πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στην δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Εμπόδια που δεν δικαιολογούνται. Μερικοί από τους πολίτες που θέλουν να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υπογράψουν. Μια μελέτη που έγινε από το τμήμα μελετών πρόσφατα επίσης αναφέρει τα σημεία αυτά και περιγράφει ε, τις διευθετήσεις αυτές ε, ότι καθιστούν την πρωτοβουλία δυσχερή στη χρήση ε, και τονίζει ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ περίπλοκο σύστημα πολλαπλών ε, συνόλων ε, προϋποθέσεων εθνικών προσωπικών δεδομένων που αποτελεί απαγόρευση για περίπου 11 εκατομμύρια πολίτες. Η αρχική πρόταση της Κομισιό είχε απαιτήσεις πιο απλές και ενιαίες για όλα τα κράτη-μέλη που θα επέτρεπαν σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία πολιτών. Λόγω της απαιτούμενης προσπάθειας θα ήταν δυσάρεστο για τους οργανωτές να μαθαίνουν αφού έχουν επιτύχει ένα εκατομμύριο υπογραφές ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να κάνει την απαιτούμενη πρόταση νομοθετική αν είχε διατυπωθεί διαφορετικά η πρωτοβουλία των πολιτών. Βεβαίως η Κομισιόν δεν πρέπει να δωρεά με τρόπο που οδηγεί σε κατηγορίες ότι προσπαθεί να ελέγξει, να χειραγωγήσει μια πρωτοβουλία θα πρέπει να κρίνει με εύλογο τρόπο ούτω ώστε να μην απορρίπτεται μια πρωτοβουλία λόγω έλλειψης πληροφοριών από πλευράς των οργανωτών σχετικά με τον νόμο, τον ευρωπαϊκό ή τις πολιτικές ή λόγω αστοχιών στη σύνταξη. Ως προς τι λογίζεται ως επιτυχία η Κομισιό δεν θα πρέπει να έχει ως μοναδικό κριτήριο ε, την νομοθετική πρόταση. Η διαδικασία ε, είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία διότι προσφέρει στους οργανωτές μια πλατφόρμα που μπορεί να προκαλέσει δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ουσία της συζήτησης είναι και το νόημα είναι ότι διαφορετικές απόψεις μπορούν να εκφραστούν, να δοθούν αιτιολογήσεις οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν αντίθεση ή υποστήριξη με διαφανή τρόπο. Η δημόσια ακρόαση σήμερα ενέχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία οι οργανωτές να συναντήσουν την Επιτροπή και να υποβάλουν τη θέση τους με παρουσία των δύο νομοθετικών ε, σωμάτων και ίσως με υπερασπιστές και αντιπάλους πρωτοβουλίας. Είναι η δημοκρατία σε δράση ε, και θα πρέπει να πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα δημόσιας συμμετοχής, πολιτικής συμμετοχής και διαφάνειας. Επιπλέον, και θα κλείσω με το σημείο αυτό, στην συνταγματική αρχιτεκτονική της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση της πολιτικού ελέγχου ε, της μιας απόφασης της Επιτροπής σχετικά με κάθε ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευχαριστώ πολύ. Ε, περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Έχουμε μαζί μας την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που έχει συστήσει μια ομάδα ad hoc και η κυρία Άνμαρη Σίγμοντ είναι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή περνάει ο χρόνος, πολλά από αυτά που είχα υπόψη μου να πω δεν θα τα πω. Ε, πρέπει να βεβαίως να σας πω ότι ασχολούμεθα εντατικά με όλα αυτά τα προβλήματα που ετέθησαν. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την ΕΟΚΕ, από την αρχή συμμετείχαμε πολύ ενεργά και επεξεργαστήκαμε πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις ε, πάνω στις πρωτοβουλίες και θεωρούμε ότι σε μία πρώτη φάση στην υποβολή και στο τρέξιμο της πρωτοβουλίας εμείς ε, ε, ρόλο έχουμε να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία, να δημιουργήσουμε ή να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν πλατφόρμες για ανταλλαγές και όλα αυτά. Σημαντικό είναι επίσης να πούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να παρακολουθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε κομμάτι μιας πρωτοβουλίας. Είμαστε δηλαδή ουδέτεροι στην παρακολούθηση της πρωτοβουλίας. Σε μια δεύτερη φάση, όταν θα έχει επιτυχία ή θα κοντεύει να ε, ολοκληρωθεί η πρωτοβουλία μπορούμε να οργανώσουμε ακροάσεις ε, για να την υποστηρίξουμε περαιτέρω. Εδώ παίζουν ρόλο οι πλατφόρμες που ανέφερα ότι πρέπει να δημιουργούνται. Πάντοτε λέγαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα καινοτόμο μέσον για τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και γι' αυτό τα εμπόδια για μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να είναι ελάχιστα. Ε, ήδη πολλές φορές το συζητήσαμε αυτό. Στην αρχή του 2011 ε, επεξεργαστήκαμε ένα φυλάδιο για την όλη διαδικασία των πρωτοβουλειών. Ε, 60.000 αντίτυπα κυκλοφόρησαν μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες. Είναι η πιο επιτυχημένη μπροσουρίτσα που ε, εκδώσαμε ποτέ. Κάθε χρόνο από τότε διοργανώνουμε τη μέρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, 13 Απριλίου θα γίνει φέτος, για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όλους. Ε, δημιουργήσαμε μια ομάδα ad hoc που την ανέφερε και η πρόεδρος, ε, είμαι εγώ ο πρόεδρος, και συζητούμε εκεί για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βοηθούμε τις πρωτοβουλίες. Είμαστε ένα help desk ε, στην παρακολούθηση αυτών των πρωτοβουλειών για να διευκολύνουμε διάφορες δυνατότητες. Επεξεργαστήκαμε κριτήρια επίσης που πρέπει να πληρούνται από τους διατυπώνονται στην, ε, τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας και μπορούμε να τα συζητούμε και σε επίπεδο και Έχουμε και με την ΕΚΑΣ μια συμφωνία ε, συνεργασίας και δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων με υλικό τεκμηρίωσης. Είναι πολύ εκτενές το υλικό αυτό και διατίθεται σε όλους τους υπεύθυνους για τις πρωτοβουλίες. Επίσης ε, δημιουργήσαμε και μια μεταφραστική υπηρεσία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσφέρει στους οργανωτές των πρωτοβουλειών να μεταφράσουν την πρωτοβουλία με τους 800 χαρακτήρες σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο ε, έβγαλε από μια μεγάλη δυσκολία τους οργανωτές των πρωτοβουλειών για το πώς θα τα διαχειριστούν όλα αυτά. Όλα αυτά τα κάνουμε σε ένα δικό μας τμήμα, το οποίο δημιουργήθηκε από την Επιτροπή ε, και που ε, αφορά την εξυπηρέτηση της κοινωνίας των πολιτών. Θέλω σύντομα να υπησέλθω συγκεκριμένα σε ένα θέμα που αναφέρθηκε και που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ακόμα και αν μια πρωτοβουλία δεν πέτυχε το στόχο της και είναι αποτυχήσα, παρόλα αυτά είναι κομμάτι ενός πολύ σημαντικού μέσου. Δηλαδή έπαιξε το ρόλο της στην επικοινωνία. Οποιοςδήποτε άρχισε μια τέτοια πρωτοβουλία βοήθησε να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος ε, για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας όπως είπε και η κυρία Μέρτς. Αν ας πούμε κάποιο, αν ένας Γερμανός, ότι ο Ισπανός έχει το ίδιο πρόβλημα, Ένας ο Αυστριακός ότι και ο Έλληνας ενδιαφέρεται για ένα παρόμοιο πρόβλημα, αρχίζει να νιώθει Ευρωπαίος. Μην υποβαθμίζουμε λοιπόν αυτές τις πρωτοβουλίες, ακόμα και αν δεν πετυχαίνουν 100%. Γιατί ε, και αυτές έχουν συμβάλει στην, εκπλή, υλοποίηση κάποιων στόχων σημαντικών. Όλα αυτά τα συζητούμε ε, και θα δούμε και στο τμήμα της επικοινωνίας μας στην Ευρωπαϊκή ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες αυτές. Ευχαριστώ. Με την κυρία Ζίγμουντ ολοκληρώνουμε την πρώτη, το πρώτο αυτό εισαγωγικό τμήμα και θα πάμε στο πρώτο πάνελ. Από όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα είναι σαφές ότι έχουμε ελλείψεις νομικής φύσεως ελλείψεις και κενά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός του υφισταμένου πλαισίου και ακριβώς η νομική προσέγγιση θα είναι η θεματική του πρώτου πάνελ. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες μαζί μας, ε, καθένας εκ των οποίων θα έχει 10 λεπτά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Jean-Luc Sauron, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris Dauphine. Κύριε καθηγητά, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ε, πρόσκληση για ένα θέμα τόσο ενδιαφέρον. Από την εκκίνηση των πρωτοβουλίων πολιτών είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο ότι πρωτοβουλίες πολιτών μια καλή ιδέα ερωτηματικό διότι θεωρούσα ότι υπήρχε ένας κίνδυνος ε, σύγκρουσης συμφέροντος για κάποιες πρωτοβουλίες πολιτών έναντι της Κομισιόν, έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν ή όχι την τάδε ή τη δίνεα πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος μας εδώ σήμερα είναι να υποστηρίξουμε την, τον ενθουσιασμό για τις ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες πολιτών, αλλά δεν συμμερίζουμε τον ενθουσιασμό σας, διότι, μάλλον την αισιοδοξία σας, διότι βλέπουμε ότι μόνο ε, δύο εξ αυτών έχουν καταφέρει να περάσουν τα διάφορα φίλτρα, αν θέλετε, τα όρια, ενώ οι υπόλοιπες απερίφθησαν σχετικά με την ε, κατανομή αρμοδιοτήτων της Κομισιόν που είναι νομικό πρόβλημα ναι αλλά δεν είναι πάντοτε απλό να καταλάβουμε πού σταματά η αρμοδιότητα του ενός και πού ξεκινά η αρμοδιότητα του άλλου. Εγώ πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα των ECI ε βρίσκεται και στην ίδια τους τη φύση και στην τοποθέτησή τους σε μια ιστορική στιγμή όπου έχουμε μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην Ευρώπη Έχουμε κάποιες ε, τάσεις που θα έπρεπε να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες και παράλληλα έχουμε την ε, ανάπτυξη αυτής της τάσεως της ε, συμμετοχικής δημοκρατίας όπου οι επιθυμίες των πολιτών βλέπονται από τους πολιτικούς ε, ταγούς και ηθήνοντες ε, με κάποια αμφιβολία. Και αυτό ισχύει και για τους ευρωπαϊκούς ε, πολιτικούς ηγέτες, τους ευρωπαίους με συγχωρείτε πολιτικούς ηγέτες. Όλα αυτά λοιπόν εγγράφονται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο επιβραδυνόμενο θα έλεγα, διότι εάν η Επιτροπή Γιούνκερ ακολουθήσει το πρόγραμμά της, εσείς δεν θα εξετάσετε παρά 20 περίπου νομοθετικές προτάσεις ανέτος; Μιλούμε για την ε, ανακατανομή και τις εργασίες, να βρούμε δηλαδή λίγη περισσότερη δουλειά για τους ε, ευρωβουλευτές. Έχουμε μία επιβράδυνση. Και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο. Διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα μεταξύ του εκτελεστικού και του νομοθετικού σώματος στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Όμως ε, το πραγματικό πρόβλημα σήμερα στην Ευρώπη, της Ευρώπης, είναι ότι πρέπει να δράσει γρήγορα και να εξασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των ε, πρωτοβουλειών ε, πολιτών, εγώ θα πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε μια προσέγγιση ατύπων κανόνων περισσότερο παρά νομικά δεσμευτικών διατάξεων διότι αυτή ακριβώς ήταν η τάση και ακριβώς τα νομικά κενά συνεχώς τονίζονται από αυτούς που διοργανώνουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Θα πω λοιπόν τα εξή δύο. Νομίζω ότι καταρχά πρέπει να υποστηρίξουμε την ομιμοποίηση των πρωτοβουλειών των Ευρωπαίων πολιτών χωρίς να υπερτονίζουμε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκού κοινοβουλίων. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα έλεγα το εξής. Όλοι έχουν κατανοήσει ότι η Κομισιόν προσπαθεί να έχει μια συνένεση σχετικά με το νομοθετικό της ε, πλαίσιο πλάνο, ορίζοντα, και διερωτώ κατά πόσον σε μια περίπτωση διαθεσμικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλιο, αν θα μπορούσαν σε ένα τέτοιο πλαίσιο να εξετάσουν είτε τις πρωτοβουλίες των πολιτών που έχουν επιτύχει, είτε και εκείνες που δεν έχουν επιτύχει. Διότι θα μπορούσε να είναι συζητήσιμο νομικά ότι σε σχέση με την ε, TTIP, για παράδειγμα, το γεγονό ότι υπήρξε μια απόρριψη εκεί θέτει ένα πραγματικό ουσιαστικότατο πολιτικό πρόβλημα διότι έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση που κινείται προς την παράλληλη κατεύθυνση της πρωτοβουλίας που η απερίφθη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τεθούν στην επανεξέταση, ε, στην αναθεώρηση του κορονομισμού είτε σε ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που θα συνοδεύει τις πρωτοβουλίες αυτές είτε από μια πανεπιστημιακή κοινότητα ή από τις συνδικαλιστικές ενώσεις ή από άλλους πολιτικούς φορείς. Οπωσδήποτε ο συνδικαλιστικός κόσμος έχει υποστηρίξει κάποιες από τις πρωτοβουλίες αυτές Αλλά δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι η συμμετοχική δημοκρατία ε, είναι, έχει φτιαχτεί για να είναι διασκεδαστική ή ευχάριστη. Τώρα βρισκόμαστε σε, έναν, σε, ε, σε μια ευρωπαϊκή κατάσταση, πλαίσιο, ε, με μια τεράστια απέτηση για ταχύτητα, για ταχεία κίνηση προς τα εμπρός. Και μιλούμε πολύ τελευταία για ηγέτες όπως τον Ματέο Ρέντσι, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Μανιουέλ Βάλς. Και προς αυτούς τους πολιτικές ηγέτες τονίζουμε συνεχώς την ανάγκη να κινηθούν γρήγορα. Και όλα αυτά τα οποία θα επιμικίνουν τη διάρκεια μιας πρωτοβουλίας θα μειώνουν την πολιτική της αποτελεσματικότητα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν από την πρωτοβουλία σε μια ιδέα πράξεως, δράσεως. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για την Κομισιόν να απορρίψει μια πρωτοβουλία πολιτών εφόσον μια τέτοια πρωτοβουλία όπως και η Λευκή Βίβλος συνοδεύεται από μια πρόταση ανάληψης δράσεως. Και μια τέτοια πρόταση, μια πρόταση οδηγίας και κανονισμού ακόμα είναι απολύτως εντός των δυνατοτήτων των πρωτοβουλίων αυτών. Χρειάζεται επίσης μια μεγαλύτερη επιφάνεια, επικοινωνιακή ικανότητα. Δεν θα ήταν υπερβολικό μία φορά το χρόνο, στα πλαίσια ενός συμβουλίου, να τίθεται στη μερίσια διάταξη η κατάσταση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών πολιτών ώστε η ψηλή πολιτική ηγεσία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο δεν θα ήταν τόσο υπερβολικό να κοιτάζει τις ανησυχίες να εξετάζει τις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες οργανωμένα και δεν θα ήταν υπερβολικό και θα έδινε πολιτική επιφάνεια σημαντική σε αυτού του είδους πρωτοβουλίες και θα έλεγα βγαίνοντας από την νομικά θέματα ότι από εσάς ευρωβουλευτές εξαρτάται να επανυπογραμμίσετε την αναγκαιότητα των πρωτοβουλειών αυτών. Είναι μια αναγκαιότητα δημοκρατική, είναι κάτι το φυσικό γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι ανισχύει τους χ ή τους ψ ή μήπως είναι μια έκφραση του, της ανησυχίας και του άγχους των πολιτικών, των ε, πολιτών με συγχωρείτε. Αλλά για, για μένα αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όσα περισσότερα μέσα δίνουμε στους πολίτες τόσο λιγότερο τα ε, χρησιμοποιούν. Και η συνολική τάση θα έλεγα πολιτικά και κοινοβουλευτικά είναι εξαιρετικά ανισχυρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ καθηγητά Σορών και τώρα ο δόκτωρ Τάμας Μόλναρ ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κορδίνου της Βουδαπέστης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμετέχοντες, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση από τους οργανωτές στην εκδήλωση αυτή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Πριν από χρόνια ήμουν και Ζιέρ, μάλιστα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που επιστρέφω με διαφορετική ιδιότητα. Ο τίτλος της παρέμβασής μου είναι η ...που πρωτοβουλίε Ευρωπαίων πολιτών, αξιολόγηση ενός πολιτικού μέσου και ο δρόμος μπροστά. Καταρχήν, να πω ορισμένα βασικά και να αναφέρω και κάποιες αντιφάσεις. Η ΠΕΠ, Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, έχει μεγάλη σημασία μέσα στις συνθήκες γιατί έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό είναι ένα συνταγματικό στοιχείο που επηρεάζει τους στόχους και τις αξίες της Ένωσης και απορρέει από αυτές. Αν δείτε υπάρχουν τα άρθρα 1, 2, 3 στις συνθήκες σχετικά με τις βασικές μας αρχές. Μετά η δημοκρατική αξίωση ε, που στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές των άρθρων 8.3 του άρθρου 8.3 και η βάση του ΣΠΕΠ εκεί εδράζεται. Οπότε είναι πολύ υψηλά στο συνταγματικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, παρά τη συνταγματική σημασία των ΠΕΠ, δεν ε, έχει επιτύχει όσα θα μπορούσε την προηγούμενη τριετία μετά την 1η Απριλίου του 2012. Κάποια στοιχεία. Αν ε, είμαι ενημερωμένος καλά, 51 ΠΕΠ έχουν προταθεί μέχρι τώρα. 31 καταχωρίστηκαν, άρα 20, δηλαδή το 40% αυτών των προτάσεων απερίφθησαν και από τις 31 δύο είχαν επιτυχία από τις καταχωρισμένες δηλαδή και είχαμε δύο ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ως απόρρια αυτών των πρωτοβουλίων αλλά καμία δεν περιλαμβάνει και νομοθετικές προτάσεις. Και το είπαν και άλλοι αυτό, ότι υπάρχει έλλειψη νομοθετικών προτάσεων μέχρι τώρα. Το επόμενο μέρος της ε, ομιλίας μου εστιάζεται σε δύο συνταγματικές επιπτώσεις. Πρώτον, η πρωτοβουλία είναι ένα εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία, όπως λέγουν κάποιοι είναι μια προσθήκη στις υφιστάμενες δομές για τις δυνατότητες παρέμβασης των πολιτών. Στην πράξη όμως ε, είμαστε μάρτυρες πολλών αβεβαιοτήτων και γραφειοκρατικών ε, ακαμψιών και αυτό το είπαν και άλλοι ομιλητές. Και αυτό το πρακτικό πρόβλημα είναι σε κάποια αντίφαση με τον κανονισμό ΠΕΠ και το προήμιό του που ζητεί μια διαδικασία, διαδικασίες απλές ε, σαφείς, ε, φιλικές προς τον χρήστη. Όμως η στάση της Επιτροπής δημιούργησε μεταξύ άλλων εμπόδια και εδώ. Άρα τώρα έχουμε ένα δίλημα. Αν συνεχιστεί η παρούσα τάση δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι συμμετοχικής δημοκρατίας και ο στόχος να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξηθεί η συμμετοχή τους να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Επίσης, ε, η δεύτερη συνταγματική ε, επιπλοκή, η απόρρια, είναι ότι η ΠΕΠ μπορεί να επηρεάζει πολύ τις κοινωτικές μεθόδους μετά την Λισαβόνα για τη λήψη των αποφάσεων. Αλλάξτε τις διαφάνειες παρακαλώ. Οπότε εδώ ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καταλήξει σε νομοθετική πρόταση, δηλαδή παραγωγή νομοθεσίας. Ε, να, αυτό είναι ένα νομικό μέσο ε, μη ενδοτικό, ε, θα είναι δεσμευτικό μετά. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια πρόταση με βάση μια νομική πράξη της Ένωσης που απαιτείται για την εφαρμογή των συνθήκων. Όμως κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτή μια, αυτό είναι ένα μέσον ε, στα χέρια των πολιτών, το οποίο είναι ενδοτικό, μη δεσμευτικό. Ε, εγώ, ε, είναι θέμα ερμηνεία. Εγώ είμαι υπέρ τη πρώτη ερμηνεία, ότι είναι δεσμευτικό, μη ενδοτικό. Ακόμα και αν δεν είναι αποτελεσματικό αυτή τη στιγμή. Οι ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζουν πολλέ φορέ ότι τα, οι μέθοδοι τις οι κοινοτικέ θα πρέπει να ε, τροποποιηθούν επί τα βελτίο και εκφράζουν την ανάγκη για μέσα που θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ε, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων, τόσο ώστε η δημοκρατική νομιμότητα, η νομιμοποίηση να ισχυροποιείται. Ε, αν δούμε τη νομιμοποίηση εισρών νεκρών, μέχρι τώρα η νομιμοποίηση εκρών ε, είχε επιτυχία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχε επιτυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ροές όμως μπορούν να βελτιωθούν μέσα από την αποτελεσματική χρήση των ΠΕΠ. Τέλος μπορούμε να ρωτήσουμε αν αυτό το αφήγημα ας πούμε είναι ο λόγος για την ε, ε, κάποια ε, ζηλόφθονη αντίδραση της Επιτροπής που δεν θέλει να δώσει όθηση στο μέσον αυτό γιατί θεωρεί ότι εμφυλοχωρεί στα δικά της στις δικές της αρμοδιότητες. Πιστεύω ότι η ΠΕΠ θα πρέπει να γίνει απόλυτα λειτουργικό μέσον που θα δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν οι πολίτες στο έργο των πολιτικών. Ε, δεν θα πρέπει βεβαίως το, η θεματική να τίθεται μόνο από τα θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τους πολίτες. Ε, θα πρέπει να ανοίξει σε νέα θέματα η δυνατότητα των ΤΕΠ, στα πλαίσια των συνθήκων, ε, αλλά ε, να οδηγήσει και σε νέα νομοθεσία. Οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να διατυπώνονται με βάση μια συγκεκριμένη λογική και την κατάλληλη νομική βάση και χρειάζονται και νομικά ξεκάθαρες προ... Ε, προτάσεις. Άρα χρειάζονται οι πρωτοβουλίες αυτές μια σοβαρή νομική υποστήριξη για να είναι αποτελεσματικότερες. Οπότε τίθεται το ερώτημα. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού στο σημείο Β ειδικότερα συνάδουν με τη διατύπωση του άρθρου 11 παράγραφος 4 γιατί το 11.4 αναφέρεται σε νομική πράξη που ε, ε, υλοποιεί τις διατάξεις ε, ο κανονισμός λέει η μια πρωτοβουλία δεν θα πρέπει προδήλως να βρίσκεται εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση ε, στο, στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να το δούμε και όταν πρόκειται για υποβολή νέου θέματος μπορούμε την ΠΕΠ να την θεωρήσουμε ως ένα μέσον που ε, ε, ε είναι προσθετικό στο 6.5 ή στο 3.5.2 που είναι η ρήτρα για την ομοφωνία. Παράδειγμα, προστασία μειονοτήτων. Αυτό είναι μία από τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη σχετική νομοθεσία ε, παράγωγη. Οι δύο μηχανισμοί ε, όμως που υπάρχουν ήδη ε, επιτρέπουν μία πρόσβαση στο θέμα. Οι βασικές διαδικασίες ε, μόνο από τα θεσμικά όργανα μπορεί να ε, ενεργοποιηθούν. Όμως πιστεύουμε ότι η δημοκρατική συμμετοχή είναι εγγύηση για τη δημοκρατική νομιμοποίηση ε, και αυτό περνάει μέσα από τις ΠΕΠ. Συμπεράσματα. Μετά από τρία χρόνια ε, είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ε, θα πρέπει να δούμε είναι νέο κεφάλαιο αυτό για τη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή θα επηρεάσει το μέσον αυτό ή θα παραμείνει μία δήλωση πίστης στους Ευρωπαίους πολίτες που συνοδεύεται με πολλές ε, ε, ψευδεστήσεις. Ένα κενό κέλυφος και ένα κέλυφος χωρίς περιεχόμενο. Η επιτυχία των ΠΕΠ θα πρέπει να ε, υποστηριχθεί. Οι στόχοι επίσης που αφορούν την πρόθεση της δημοκρατίας θα πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ. Θα πρέπει να δούμε και τι απόφαση θα λάβει το δικαστήριο μετά από την εκδίκαση των υποθέσεων. Ε, σίγουρα μας περιμένει ακόμη πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Dr. Molnar. Ευχαριστώ, Δόκτωρα Μόλναρ. Και τώρα πηγαίνουμε στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, στον καθηγητή Φιλίπ Πουαριέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την πρόσκληση από τις δύο επίτροπες εγώ για την δική μου παρουσίαση για την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών έχω δύο, τρεις άξονες. Τρεις άξονες. Πρώτα απ' όλα το θέμα της αντίληψης και της πρακτικής της δημοκρατίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διότι έχουμε πέντε πολιτικά συστήματα με αντιλήψεις της δημοκρατίας δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ΠΕΠ αν δεν την τοποθετήσουμε σε ένα πλαίσιο επαναπροσδισμού των σχέσεων της δημοκρατίας και της νομιμότητας στην Ένωση και στα κράτη. Και μετά θα ασχοληθώ με τρόπο επικριτικό την ΠΕΠ και όπως και οι συνάδελφοί μου θα αναφερθώ σε ορισμένες πρόπτικες. Όταν κοιτάζουμε τις διάφορες αντιλήψεις δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σας παρακαλώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ανταγωνιστικές και συμπληρωματικές. Περνάμε γρήγορα τις διαφάνειες, διότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Υπάρχουν πέντε μεγάλες αντιλήψεις που είναι ε, συμπληρωματικές και καμιά φορά συνεργάζονται. Η διαδικαστική των κανόνων, η λυτρωτική και ένα μέρος των πρωτοβουλειών προέρχονται από την οικονομική και ελιτίστικη δημοκρατία εκτός των τριών. Αν δούμε στο επίπεδο της πρακτικής άλλες διαφάνειας της δημοκρατίας υπάρχει μια ένταση δημιουργική και μια σύγχυση στις πρωτοβουλίες των ε, κοινοβουλίων και των ατόμων ανάμεσα στην συμμετοχική, στην διαβουλευτική δημοκρατία, στην λογική δημοκρατία και περνάμε αμέσως στην συμμετοχική δημοκρατία, διότι δεν θα έχουμε χρόνο. Σχετικά με την συμμετοχική δημοκρατία υπάρχουν τρία στοιχεία που ξεχνούμε στις αναλύσεις μας. Πρώτον, εξορισμού οι δημοκρατίες αυτές έχουν ένα μοραλισμό πολιτών και αυτές οι πρωτοβουλίες που απορρίφθηκαν ή δεν έγιναν δεκτές εξαρτώνται κυρίως από αυτήν την κατηγορία. Δεύτερο στοιχείο, η συμμετοχική δημοκρατία ε, ενέχει ε, την αρχή ε, της συνεκπώνησης της νομοθετικής και εδώ είμαστε μακριά από την ΠΕΠ την Ευρωπαϊκή. Και τρίτο στοιχείο είναι η συνυπευθυνότητα και εδώ δεν είμαστε καθόλου σε αυτό το πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις αντιλήψεις των διαφόρων δημοκρατιών, ας περάσουμε τώρα ε, στην επαναπροσδιορισμό της σχέσης ε, μεταξύ δημοκρατίας και νομιμότητος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Είναι μια έρευνα περίπου 30 ετών, δεν χρησιμοποιώ το παρόμετρο, αλλά χρησιμοποιώ άλλες βάσεις που διαπιστώνουν μια υποχώρηση συνεχή της νομιμότητας στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Πώς να βρούμε λοιπόν τα μέσα και αποκρίνεται σε αυτά τις απαιτήσει. Θα περάσουμε στις άλλες διαφάνειες και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άλλες έρευνες του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ε, σε συντονισμό με πανεπιστήμια βλέπουμε ότι οι πολίτες ζητούν μηχανισμούς διαφάνειας, τους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων ε, και εκπόνηση μηχανισμών συμμετοχικής δημοκρατίας. Ταυτόχρονα έχουμε μια κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς τα κόμματα περνάμε και στις άλλες διαφάνειες και στην ε, έλλειψη υποχώρηση, στην προσχώρηση και στράτευση σε πολιτικά κόμματα. Βλέπουμε επιθυμία κυρίως στην ε, Γερμανία, πάνω από 65% θέλουν μέσα ε, στο επίπεδο του κράτους, της περιφέρειας και της Ένωσης για συμμετοχική δημοκρατία. Πρέπει να αποκατασταθεί. Και τώρα ερχόμαστε στην ίδια την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτικών και στις ε, πρόπτικες της. Άρθρο 10. Εδώ θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Θα ενδιαφερθώ για τη συνθήκη και για τον κανονισμό. Στο άρθρο 10 της συνθήκης έχουμε τις τρεις αρχές της ε, δημοκρατίας της συμμετοχικής και αντιπροσωπευτική Ο λειτουργία της Ένωσης βασίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στην δημοκρατική ζωή, αλλά έχουμε και την μεσολάβηση διαμέσου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Στο άρθρο 11, επόμενη διαφάνεια, έχουμε ένα δίπολο αντιπροσώπευσης της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης. Έναν διάλογο ε, μη δεσμευτικό της με την αρχή της δαφάνειας ανάμεσα στα στοιχεία. Όταν μιλάω για δίπολο είναι ότι οι συνθήκες αφήνουν ένα χώρο, μια θέση για τους πολίτες αλλά και για τις οργανώσεις οι οποίες διαμεσολαβούν για να αντιπροσωπεύσουν τα συμφέροντα των πολιτών. Θα αφήσουμε και τα άλλα άρθρα την διαδικασία και ερχόμαστε σε στοιχεία ανάλυσης του κανονισμού ως έχει σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την αρχή της κεντρικότητας της Κομισιόν σε αυτών των κανονισμών. Είναι η Κομισιόν η οποία είναι ο βασικός παράγων. Μετά υπάρχει μια αρχή ενύπαρξης που αφήνεται στους πολίτες, ένα δικαίωμα για τους πολίτες που μπορούν να οργανώνονται μόνοι τους χωρίς τις οργανώσεις που εξαρτώνται από ομάδες συμφερόντων. Αυτό είναι μάλλον ε, μια διαπίστωση ε, πολιτολογίας συνήθως οργανώνονται διαμέσου των ΜΚΟ, των συνδικότων. Να πούμε ότι υπάρχουν μια αυθυπαρξία οι πολίτες αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει θέση ε, λοιπόν για τους ίδιους τους πολίτες, διότι τα κόμματα τα πολιτικά καμιά φορά δεν έχουν ε, την οργάνωση ε, για να οργανώσουν μια πρωτοβουλία. Υπάρχει αναλογικότητα, υπάρχει επικουρικότητα για τα κράτη-μέλη και η Κομισιό παρουσιάζει στην διατύπωση του κανονισμού και αυτό είναι ενδιαφέρον, τα πορίσματα τα νόμικα αλλά και πορίσματα πολιτικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο πολιτικό που θα πρέπει να συζητηθεί ή να απορριφθεί και υπάρχουν ε, και όροι ε, διαφάνειας και εξωτερικής συμβολής παρόμοια με αυτήν των κομμάτων των ευρωπαϊκών των πολιτικών. Αν δούμε τις επόμενες διαφάνειες, διότι ήδη αναφέρθηκαν οι συναδελφοί μου στην απόρριψη Ποια είναι τα όρια τα οποία ήδη ανέφερα. Πρώτο όριο η ιδέα ότι μια κοινωνία πολιτών αποτελείται από άτομα, ενώ αποτελείται από ομάδες συμφερόντων συνήθως. Πρέπει λοιπόν πώς να συνδέσουμε καλύτερα τις ομάδες συμφερόντων, τις ΜΚΟ, συνδικάτα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών. Η πρότασης δεν πρέπει να είναι αντίθετες προς τις αξίες της Ένωσης. Αυτό είναι ένα πλαίσιο κανόνων και προτύπων που είναι ενδιαφέρον, αλλά κάπως περιορίζει την πρωτοβουλία και ως προς την ουσία ε, της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε εκεί ότι έχουμε τη διακυβέρνηση, την οικονομική και την ενιαία εσωτερική αγορά. Ε, ο έλεγχος εξ ε, επιτρέπεται σε σχέση με την σκοπιμότητα εξ να αποφασίζει όχι να δώσει συνέχεια είναι κάτι το σημαντικό αυτό ο έλεγχος. Πρώτα απ' όλα διαμέσου εμπειριών στο επίπεδο των εθνικών κοινοβουλίων ή των περιφερειακών κοινοβουλίων αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον θα ήταν να σκεφτούμε στην αρχή στην αρχή μιας θητείας να υπάρξουν θέματα και κατάλογοι που να αντιστοιχούν ε, στις εντολές που έχουν δοθεί και όπου οι πρωτοβουλίες οι ευρωπαϊκές θα μπορούσαν να λάβουν χώρα. Δεύτερο στοιχείο σε σχέση με τα εθνικά ή περιφερειακά ε, κοινοβούλια εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν ευκταίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να τίθεται στο επίκεντρο της ε, τεχνικής και νομικής διαδικασίας ούτω ώστε να ενισχύεται και η νομιμότητα που ανέφερε ο συνάδελφος Σωρό. Τρίτον, η, η πρωτοβουλία αν είναι δεκτή στους κανόνες θα έπρεπε να είναι ένα από τα στοιχεία συμμετοχικής δημοκρατίας δεσμευτικό. Ένα από τα στοιχεία τα δεσμευτικά σε μια ατζέντα νομοθετική. Είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, Ιδανιώ το μέσο αυτό χάνει την εγκυρότητα για τους πολίτες. Τέλος, Όσο προς την δημοσιοποίηση είναι ενδιαφέρον η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών να συνδέεται με τις πρωτοβουλίες των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων για να ε, αποφύγουμε να υπάρχουν ε, αντιφάσεις ή επικάλυψη και ελευθερό στοιχείο πολύ σημαντικό τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στην δημόσια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν ε, να έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν τουλάχιστον μια πρωτοβουλία στη θητεία τους και έτσι ε, θα μπορούσαν οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, τελευταίο στοιχείο, οι ομάδες συμφερόντων θα έπρεπε επίσης να συμμετέχουν. Θα έπρεπε λοιπόν να τα τοποθετήσουμε αυτά στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών δεν θα έπρεπε να συνδυάζονται και τα τρία στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον ομίλητη. Έχουμε 15 με 20 λεπτά τώρα, ανάλογα με το πόσοι από εσάς επιθυμούν να έχουν το λόγο. Θα προσπαθήσω να σημειώσω τα ονόματά σας. Παρακαλώ να έχετε υπομονή. Θα έχουμε δύο λεπτά ανά άτομο για να έχουμε και κάποιο ελάχιστο χρόνο απαντήσεων. Ο κύριος Ογιασδόσκη. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που σε αυτό το πρώτο μέρος της ε, συζήτησης έλειψε ένας εκπρόσωπος της One of Us, της πιο δημοφιλούς ε, πρωτοβουλίας με τις περισσότερες υπογραφίες ε, και με στήριξη από 20 διαφορετικές χώρες. Ήταν σίγουρα η δημοφιλέστερη από τις πρωτοβουλίες. Ε, θα μου άρεσε κάποιος που εκπροσωπεί τη One of Us να ήταν παρόν. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι το εξή Η Κομισιόν μπορεί να απορρίψει μια λαϊκή πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία των πολιτών που υπακούει, συμμορφούνται προς όλους τους τυπικούς κανόνες. Ερωτηματικό. Ο Επίτροπος Τίμερμανς μας λέει για ανοιχτό πολιτικό διάλογο και για διαθεσιμότητα της Κομισιόν, αλλά τελικά θα υπάρξει κάποιος περιορισμός σχετικά με, το, με τον τρόπο με τον οποίο θα είναι ελεύθερη να αποφασίζει η Κομισιόν. Σχετικά δηλαδή με την αποδοχή αυτών των, την σημείωση αυτών των σημαντικών ετοιμάτων των πολιτών. Η περίπτωση της One of Us είναι πραγματικά χαρακτηριστική διότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ε, να μετατραπεί αυτό το δικαίωμα, το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών σε επιστημονική φαντασία στην πραγματικότητα. Εφόσον η Κομισιόν αγνοεί τις πρωτοβουλίες αυτές. Ελπίζω λοιπόν ο Επίτροπος και η Κομισιόν γενικά να οδηγηθεί σε μια αλλαγή και σε ένα περιορισμό του τρόπου με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις Νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να είναι ελεύθερη να λαμβάνει αρνητική απόφαση μόνο σε εξαιρετικές αποφάσεις και υπό συγκεκριμένου κανόνες. Αναφέρθηκαν τώρα και οι καθηγητές ε, για την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Ο κύριος ε, ο καθηγητής Παγιέ μας είπε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα όπως αντίθετα σημαίνει στην Γαλλία όπου μετά τη μεταρρύθμιση του 2008 μπορούν να υποβάλουν νομοθετική πρόταση συγκεκριμένοι οι πολίτες. Μάλιστα, εντάξει, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συνάδει προς την κατεύθυνση την οποία σημειώνα προηγουμένως. Δεν μπορεί η Κομισιόν να αποφασίζει όπως θέλει εκείνη. Επομένως την επιχειρηματολογία του καθηγητή την θεωρώ ακριβώς ε, παράλληλη προς, την, ε, το δικό μου αίτημα να περιορίσουμε αυτήν την αυθαιρεσία της Κομισιόν. Ε, δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τα δύο λεπτά, λέει η Πρόεδρος, διότι δεν θα έχουμε καθόλου καιρό. Γιόλα είναι δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, τρεις πρωτοβουλίες είχα υποβάλει. Η μία είχε επιτυχία, οι άλλες απέτυχαν και είδα τις δυσκολίες και τα ελλείμματα του μέσου. Πάντως όλοι συμφωνούμε ότι είναι εκ των όνων κάνευ το μέσο αυτό για τους πολίτες και τη συμμετοχική δημοκρατία που χρειαζόμαστε τόσο κατεπηγόντως επειδή φαίνεται να είναι μακριά η Ένωση από τους πολίτες. Άκουσα τις τρεις ομιλίες, πολύ ενδιαφέρουσες. Στο μέλλον το εύρος της πρωτοβουλίας των πολιτών πρέπει να ε, γίνει ακόμη μεγαλύτερο και να αναβαθμιστεί η νομιμοποίηση. Στηρίζω αυτά που ελέγχθησαν οι πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να περιορίζονται στις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να επεκτείνονται και στην αρμοδιότητα που καλύπτουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, που είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως παράγοντα που δρά αυτοβούλος και μπορεί και να νομοθετεί μάλιστα. Δηλαδή πάει πολύ πιο πέρα από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα υπάρχουν πολλά θέματα ε, στα οποία πρέπει να, τα οποία πρέπει να ανοίξουν για τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Ε, επίσης πρέπει να αναβαθμιστεί η νομιμοποίηση, όπως είπε και ο καθηγητής Σωρών. Εσείς κυρία Κάουφμαν είσαστε εισηγήτρια ε, όταν ε, ε, αναφερθήκαμε σε μια πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προϋπέθεται συμβαστική λύση με το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο όμως ε, έχει και έμεσο δικαίωμα νομοθετικών πρωτοβουλειών το οποίο το αποκτήσαμε μετά από μάχη πριν από 10 χρόνια. Η πρωτοβουλία των πολιτών δεν πρέπει να απευθύνεται λοιπόν μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τουλάχιστον και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην πω και το, Ευρωπαϊκό, και το Συμβούλιο των Υπουργών γιατί και εκεί υπάρχουν τομεί όπου λαμβάνει νομοθετικές ε, ε, αποφάσεις στο Συμβούλιο. Εμείς τα παρακολουθήσαμε όλα αυτά και μέσα από τη συνέλευση, μέσω της Επιτροπής ΑΦΚΟ και τώρα μέχρι την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα Ουγγρικά. Κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ για την τωρινή πρωτοβουλία, για την εκδήλωση. Ως Ευρωπαίος Βουλευτής ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι γίνονται τόσες προσπάθειες για τις ΠΕΠ. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρει μεγάλη ευθύνη, έχει αναλάβει μεγάλη ευθύνη. Ε, εμείς θα πρέπει να δώσουμε γνωμοδότηση και σύσταση για τη βελτίωση του συστήματος. Η Επιτροπή Αναφορών θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και η συγητής. Ε, η συζήτηση μέχρι τώρα έδειξε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ε, για το κλίμα χρειάζεται ένα σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να βελτιωθούν και οι μηχανισμοί μείωση τη γραφειοκρατία. Οι διαδικασίε πρέπει να γίνουν λιγότερο γραφειοκρατικέ, γιατί ακούσαμε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Και υπάρχει και ένα τρίτο τομέα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί εδώ. Πρέπει το σύστημα να αλλάξει ούτω ώστε να μην λαμβάνει την τελική απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών. Χρειάζεται και, ένας, ε, και ένα άλλο θεσμικό όργανο που θα συναποφασίζει και θα ενέχεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος που εκπροσώπησε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Ε, πάνω εκεί πρέπει να δουλέψουμε. Κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντική ημέρα και για μένα. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τόσο πολλούς ειδικού για το θέμα και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη διότι ε, έχουμε αυτή την τριετή διορία στον κανονισμό και έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα μετά τις πρώτες εμπειρίες να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του κανονισμού. Το μέσο αυτό Πώς το διαχειρίστηκαν οι πολίτες, πώς το κρίνουν, πώς ε, λειτουργήσε, έδρασε, τι πολιτικό ρόλο έχει. Αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία που αναφέρθηκε και εδώ και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Πιστεύω ότι ακόμα είμαστε σε ένα πειραματικό στάδιο. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι κάτι διεθνώς μοναδικό. Εμείς την θεσμοθετήσαμε και μετά από τρία χρόνια πρέπει να δούμε πώς λειτουργήσε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν προς όλους. Ακούσαμε πολλές προτάσεις για αλλαγές και παρακαλώ τη γραμματεία μετά την ακρόαση να καταγράψει τα θέματα αυτά που είναι τόσο πολλά και διαφορετικά γιατί όλοι φέρουμε ευθύνη από κοινού. Οι παρατηρήσεις του Αντιπροέδρου Τίμερμανς ε, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικές. Χαίρομαι διότι με μεγάλη σοβαρότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα προχωρήσει στην υποβολή της έκθεσής της και εμείς ως Κοινοβούλιο πάνω σε αυτή τη βάση θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, τι συνέχεια θα δώσουμε στην ε, δυνατότητα αυτή για ΠΕΠ. Θεωρώ μετά από αυτά που άκουσα μέχρι τώρα ότι ένας θα είναι ο στόχος, ο κύριος, να γίνει η επεξεργασία του κανονισμού, αναθεώρησή του και να δούμε πώς θα γίνει απλούστερο το μέσον ε, που θα χρησιμοποιείται από τους πολίτες. Αν αυτό είναι ο στόχος μας, έχω και μία παράκληση. Χρειαζόμαστε το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και όπως είπε και ο Γιώ Λάινεν πιο πριν, ε, δυστυχώς ε, έχουμε πολλή γραφειοκρατία. Σκεφτείτε τους διαφορετικούς καταλόγους για τη συλλογή υπογραφών κλπ. Και πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο γιατί χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη. Όλοι τα κράτη-μέλη μας θα πρέπει έγκαιρα να αποκαταστήσουμε τις απαραίτητες επαφές ούτως ώστε γρήγορα να βελτιωθεί η δυνατότητα που έχουμε για ΠΕΠ. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι βεβαίως δεν είμαστε μόνο εδώ, το Συμβούλιο δεν είναι μόνο εδώ για να ακούει αλλά και για να για να μιλάει αλλά και για να ακούει. Uh, I ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο, ο καθηγητής ε, Σογό μίλησε για μια σύγκρουση νομιμοποίησης. Και επομένως πού είναι ο βασικός κανόνας. Υπάρχει μια ιεραρχία νομιμοποίησης. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η προσέγγιση τελικά που ακολουθούμε. Ανεξαρτήτως του που οδηγεί και αυτή εδώ η συνάντηση και γενικά η έκθεση. Και συμφωνώ ότι ε, αυτό είναι το βασικό που πρέπει να μας ε, απασχολήσει και εγώ ως συζητητής αυτό θα θεωρήσω ότι είναι η βασική γραμμή. Ευχαριστώ. Richard Corbett σας ευχαριστώ. Πάντα υπήρξα επιφυλακτικός ε, σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτών για τον εξή λόγο. Εάν κάτι είναι καλή ιδέα, γιατί χρειάζεται ένα εκατομμύριο ελεγμένες υπογραφές να υποβληθεί στην Κομισιόν. Δεν θα έπρεπε να μπορεί οποιαδήποτε μικρή ομάδα να υποβάλει μια καλή ιδέα. Και αν κάποιος είναι σε θέση να έχει ένα εκατομμύριο ελεγμένες υπογραφές και υπάρχει επομένως μια δημόσια στήριξη, σίγουρα θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται στο πολιτικό γίγνεσθε, στο πολιτικό γήπεδο. Είναι δυνατόν κανέν, καμία, κανένας μη όμικρον ή κανένας άλλος φορέας να μην έχει ήδη θίξει το θέμα αυτό. Και επομένως υπό την έννοια αυτή έχουμε δημιουργήσει ένα εμπόδιο. Και δείτε το διαφορετικά. Αν κάποιος πιάσει 990.000 υπογραφές, αλλά η Κομισιόν πει, λοιπόν όχι, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Τότε τι θα πει η Κομισιόν. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί δεν έπιασε 10.000 υπογραφές ακόμα. Δεν νομίζω. Επομένως, κατά την άποψή μου πρέπει τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο απλά. Η συνθήκη δεν πρόκειται να αλλάξει. Ας την κάνουμε να λειτουργήσει καλύτερα ίσως. Και σε πρώτη... Ως πρώτο βήμα δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την Κομισιόν να αποδέχεται οποιαδήποτε ιδέα φαίνεται ότι θα μπορούσε να μαζέψει ένα εκατομμύριο υπογραφέ, χωρί να χρειάζονται όλε αυτέ οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε ελέγχου, κόντρα ελέγχου κτλ. των υπογραφών. Γιατί αν κάποιο φτάσει στι 800 ή 900 δεν αξίζει να δώσουμε μια απάντηση ακόμα και αν η απάντηση είναι αρνητική. Αντί να πάμε να ψάξουμε στα συρτάρια της γραφειοκρατίας να δούμε αν κατά πόσον ελέγχθηκαν σωστά οι υπογραφές, αν καταχωρίστηκαν σωστά τα διαβατήρια, οι αστυνομικέ ταυτότητες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εφόσον κάτι φαίνεται ότι μαζεύει σημαντική στήριξη, ας μην κολλάμε σε αυτά τα νούμερα. Ναι, Είχαμε πολλές ε, περιπτώσεις ε, ε, των καλύτερων κοινοβουλίων και των μεγαλύτερων κοινοβουλίων στον κόσμο που έχουν περάσει πρωτοβουλίες όχι τόσο ευφύς. Δεν είναι πάντοτε εγγύηση δηλαδή αυτό που λέτε. Τέλος πάντων, ανόητο σχόλιο εγώ τώρα κάνω, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Κάμπρας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα είναι η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών ως μέσο να γίνει πιο γνωστό και πιο διαφανές και αναφέρομαι σε τρία σημεία που δεν είναι νέα αλλά που είναι νομίζω λογικά και μπορούν να βοηθήσουν. Οι πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να έχουν υποδομή στήριξης, νομικές συμβουλές και καθοδήγηση για την απαραίτητη εκστρατεία και πρόθεση η ικανότητα των οργανωτών ε, ενέχει ορισμένους κινδύνους. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διεθνική νομική οντότητα ε, για την ε, Επιτροπή των Πολιτών. Τρίτον, σχετικά με τις απαιτήσει ως προς τα στοιχεία, τα δεδομένα, θα πρέπει να απλουστεθούν σε όλα τα κράτη-μέλη και να απορρίψουν, να αποκλείσουν ε, τον αριθμό ταυτότητας ε, που ε, υπάρχει. Θα πρέπει οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας θα πρέπει να δίνουν το όνομα, τη διεύθυνση και την εθνικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τους τρεις ομιλητές Ας αρχίσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Πουάριε. Είναι το Λουξεμβούργο έτοιμο. Το Λουξεμβούργο δεν είναι έτοιμο. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις είναι πάρα πολύ επικοδομητικές και συμπληρώνουν ε, την παρουσία σήμως. Μην νομίζετε ότι είναι αγένεια εκ μέρους μας που απαντάω έτσι. Είναι καλύτερα όμως νομίζω. Ο καθηγητής κύριος Μόλναρ. Ναι, άκουσα τις διάφορες παρεμβάσεις. Συμφωνώ με πολλές συγκεκριμένες προτάσεις που έγιναν από ευρωβουλευτές λόγω της έλλειψης χρόνου, όμως δεν μπορώ να κάνω συγκεκριμένα σχόλια σχετικά με τις παρεμβάσεις. Ε, και επειδή δεν μου ζητήθηκε να δώσω τέτοια σχόλια, θα δώσω το λόγο σε άλλους που βρίσκονται εδώ. Ρωτηθήκατε ρητά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σημείωσα ότι έπρεπε να απαντήσω. Νομίζω ότι οι 15 τελευταίες μέρες δείχνουν ότι υπάρχει στην Ευρώπη μια σύγκρουση νομιμοτήτων ανάμεσα στους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, τον λαό της Ελλάδας και το Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Υπάρχει μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση και στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει ένας κατατεμαχισμός εξουσιών, ένας πολλαπλασιασμός εξουσιών, ένα μικρό κομμάτι στους πολίτες, ένα μικρό κομμάτι εδώ εκεί, ενώ δεν αλλάζει το σύστημα το θεσμικό στις Βρυξέλλες. Ενώ λοιπόν έχουμε αντίθετες δυνάμεις υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι ε, είναι σημαντικό στην μεταρρύθμιση ε, ε, και την αναμόρφωση του κανονισμού να υπάρξει μια, μια συνεργασία, τα εθνικά κοινοβούλια που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν. Οι, Βρυξέλλες προσπαθούν να παρακάμψουν τις, τους εθνικούς θεσμούς, τις εθνικές δομές προς όφελός της η Επιτροπή. Αυτό είναι άδικο για τις Βρυξέλλες, αλλά πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Να υπάρξει λοιπόν ε, μια ενορχίστρωση των νομιμοτήτων, μια συνεργασία ε, και μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής ε, και είδαμε στις παρεμβάσεις ότι όταν υπάρχει μια πρωτοβουλία που προωθήθηκε με τρόπο σημαντικό στο ΠΕΙΠΕ ε, και δεν υπάρχει πρόβλημα νομικό, βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι που δεν προχωράει καλά. Θα πρέπει λοιπόν οι τρεις Συμβούλιο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο να βρούνε το πολιτικό πλαίσιο και το, να δώσουν απάντηση στους πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, τελειώσαμε με το πρώτο πάνελ, αλλά θέλουμε ακόμη να πούμε κάτι Νομίζω ότι βρισκόμαστε τώρα στην ε, διαδικασία όπου η Επιτροπή δουλεύει για το μέλλον και προσπαθεί να δει την ε, κανονισμό ως προς τα κενά ε, της ελλείψης και ως προς την πολιτική της σημασία πράγματι αποδίδει ως πολιτική νομιμότητα αλλά επίσης εμείς θέλουμε τα σχόλιά σας εδώ στο Κοινοβούλιο διότι οι δύο επιτροπές έχουν να κάνουν έκθεση. Γι' αυτό χαιρόμαστε ε, για την, ε, τη σχόλιά σας. Εσείς προέρχεστε από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά μας ανοίγετε νέες προοπτικές για τα θέματα που σχετίζονται με την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε βεβαίως τις γραπτές σας ε, παρουσιάσεις ή θα τις έχουμε. Συνεπώς όποιος ενδιαφέρεται μπορεί αργότερα να τις ε, λάβει από το ε, Κοινοβούλιο. Ε, δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τους ευρωβουλευτές, τους εκλεγμένους, γιατί ασχολούνται με το βασικό στοιχείο της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών και διευρύνουν την εμβέλεια αυτής της δυνατότητας. Είναι τιμή να είναι κανείς εκλεγμένο μέλος του Κοινοβουλίου. Το προηγούμενο πάνελ ήταν για τα νομικά θέματα. Τώρα προχωρούμε στο δεύτερο πάνελ, η δεύτερη συνεδρία, που θα επικεντρωθεί στις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή των πρωτοβουλειών Ευρωπαίων πολιτών. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω τους εξής ομιλητές. Πρώτον, τον κύριο Κάρστεν Μπέρ, Γενικό Συντονιστή της εκστρατείας ΠΕΠ, τον κύριο Φρανσίσκο Πόλο, ο οποίος είναι διευθυντής της χώρας στην Ισπανία και διευθυντής της ε, Παγκόσμιας Διεύρυνσης στη Μαδρίτη ε, από την πλατφόρμα change.org, την κυρία δόκτωρα Σουζάνα Ντελρίο Βιλάρ, που είναι συγγραφέας και διευθύντρια του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναβάθμισης Ευρώπης. Πολύ φιλόδοξος στόχος. Δεκά λεπτά έχετε ο καθένας και παρακαλώ να σεβαστείτε αυτό το χρόνο ομιλίας. Μετά θα ακολουθήσει συζήτηση με ρωτήσεις απαντήσεις. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω γιατί συνήθως οι πολιτικοί μακρηγορούν άμα βρεθούν μπροστά σε ανοιχτό μικρόφωνο. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό, τουλάχιστον όχι τώρα. Ανταυτού δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπέρκ για 10 λεπτά περίπου. Ευχαριστώ πολύ. Τις διαφάνειες παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι μέλη των Επιτροπών Αύκο και Πέτη, ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης που είναι πάρα πολύ επίκαιρη τώρα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση να είμαι ομιλητής. Επόμενο, επόμενη διαφάνεια. Είναι τιμή μου που εκπροσωπώ την ECI Campaign, την, καμπάνια PEP, e που εδώ και 10 χρόνια εργάστηκε για αποτελεσματικό δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλία των πολιτών της Ευρώπης. Η PEP e έχει πολλούς γονείς όμως. Είναι παιδί μεγάλης οικογένειας. Πολλοί γονείς παρευρίσκονται εδώ σήμερα. Θα θυμάστε ότι ποτέ δεν την ήθελαν την ΠΕΠ οι κυβερνήσεις. Εσείς όμως εδώ οι βουλευτές μαζί με οργανώσει της κοινωνίας των πολιτών ε, εργαστήκατε ούτως ώστε να ενταχθεί στην ε, συνέλευση για τη σύμβαση για το μέλλον της Ευρώπης του 2002. Κύριε Στίμαρσον είναι εδώ, κυρία Χουίμπνερ, κυρία Κάουφμαν, ε, κύριος Μπρόκ, κύριος Λαμασούρ και οι εισηγητές Χέφνερ Μόρις. Είναι πολύ καλό ότι ε, αυτή η κοινότητα παλιών και νέων μελών συνεχίζει να υπάρχει γιατί εμείς ε, είμαστε ένας έμπιστος εταίρος ε, περισσότερων από 25 καμπάνιες ΠΕΠ. Ε, σημειώσαμε τις αλλαγές που ε, υπήρξαν. Επίσης δημοσιεύσαμε μια έκθεση, μια γνώμη σχετικά με την έκθεση του 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΠΕΠ Τώρα μετά από τρία χρόνια θα πρέπει να αξιολογήσουμε το σημείο καμπή στο οποίο βρισκόμαστε, να λάβουμε δράση. Όλοι μας είπαν, μέχρι τώρα οι ομιλητές είπαν ότι έχει πολύ μοιραία ασφάλματα ο κανονισμός και οι οργανωτές των ΠΕΠ ε, καλούνται να συμμορφωθούν με άσκοπες διαδικασίες επαχθής αν δεν πάμε τώρα για απλοποίηση και βελτίωση του κανονισμού ΠΕΠ, η διαδικασία θα σταματήσει, δεν θα λειτουργείται πια και θα είναι μια υπόσχεση κενή περιεχομένου. Μία ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πολλοί πιστεύουν ότι έχασε το δρόμο της. Βλέπετε πόσοι ευρωσκεπτικοί στές υπάρχουν, πόσοι ε, αντιευρωπαίοι που εξελέγησαν και εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί με τους πολίτες, όχι ερήμην τους. Πρέπει λοιπόν τώρα να ξεδιπλώσει το δυναμικό που έχει και η πρωτοβουλία το μέσον ΠΕΠ. Είναι μοναδική ευκαιρία για όλους μας. Ας φροντίσουμε να γίνει το σωστό. Πώς κρίνουμε λοιπόν αυτό το μέσον ε, υπερεθνικής συμμετοχικής διαδικασίας ε, ποια είναι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε για να το αξιολογήσουμε ένα σημαντικό κριτήριο είναι να βεβαιωθούμε ότι οι ΠΕΠ χρησιμοποιούνται γίνονται επόμενο βλέπουμε σε αυτή την διαφάνεια την εξέλιξη των αριθμών αρχίζοντας το 2012 μέχρι το, το, τέλος του 2014. Είχαμε περισσότερες από 50 ΠΕΠ καταχωρισμένες, ε, ε, υποβληθήσεις. Μόνο 26 καταχωρίστηκαν, ε, τρεις υπέτυχαν να συγκεντρώσουν το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Το 2013 είχαμε μια κορυφή και μετά καθοδική πορεία. Δεν ε, γίνεται τίποτε πια. Επόμενο η διαφάνεια δεν λειτουργεί πια αυτή η δυνατότητα και αυτό το δείχνουν και οι διαφάνειες. Και εδώ βλέπετε το 2012-2013 κορύφωση αριθμού υπογραφών, τώρα είμαστε κοντά στο μηδέν. Αυτό το μέσον δεν αξιοποιείται πια από τους πολίτες. Γιατί Ξέρουμε από εθνικές πρωτοβουλίες ε, πολιτών ότι μόνο αυτές που είναι σχεδιασμένες με φιλικό τρόπο προς τους πολίτες και επηρεάζουν τις ε, σχετικές πολιτικές, μόνο αυτές ε, οι πρωτοβουλίες χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας τώρα με τον επανέλεγχο του κανονισμού και την αναθεώρησή του. Γι' αυτό ε, συμφωνήθηκε στο προήμιο του κανονισμού ότι οι διαδικασίες και παραθέτω τώρα οι διαδικασίες πρέπει και οι, όροι πρέπει να είναι ε, σαφείς, απλές, φιλικές προς το χρήστη, αναλογικές προς τη φύση της πρωτοβουλίας των πολιτών για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή από τους πολίτες και για να γίνει πιο προσπελάσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι όμως απλές, σαφείς και φιλικές προς το χρήστη και δύσκολα χρησιμοποιείται το μέσο ΠΕΠ για την, ε, ως μέσο άμεσης δημοκρατίας. Δεν αλλάζει όμως το, τους νόμους, ε, δεν λαμβάνει αποφάσεις η διαδικασία ΠΕΠ, δεν απαιτεί ανάληψη δράσης, μόνο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την προσθήκη ενός θέματος στο, στην ατζέντα της. Αυτό, ε, αυτό είναι υπερεθνικό, επίσης έχει υπερεθνικό χαρακτήρα, δηλαδή ε, είναι δύσκολο να εντάξουμε πολίτες που μιλούν 22 διαφορετικές γλώσσες 26 χώρες. Πώς θα μεταρρυθμίσουμε λοιπόν το ΠΕΠ όταν γίνει η επανεξέταση. Πώς θα ε, μεταρρυθμίσουμε το ΠΕΠ. Εμείς ε, παρατηρούμε ε, μετά από τις συζητήσεις και ζημώσεις που έγιναν ότι αναδύονται τρεις ε, τομείς. Πρώτον, για αλλαγή. Η καταχώρηση πρέπει να γίνει με λιγότερο περιοριστικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίρνει στα σοβαρά τις επιτυχίες ΠΕΠ και οι προϋποθέσεις για τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τροποποιηθούν, δηλαδή να μην χρειάζεται αριθμός ταυτότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή de facto περιόριζε την ελευθερία του λόγου, αυτό παρατηρήσαμε, όταν απορρίπτει περίπου το 50% από την καταχώρηση. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ μη παραδεκτού και αποτυχίας ο, αν δούμε τις πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο. Και όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κάνουμε. Δεν αφήνουμε τους πολίτες μας να μιλήσουν. Και ε, λέμε, και το είπε και ο Γιώργο Λάινεν, πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής. Ε, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει αλλαγές στη συνθήκη και οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ΟΠΕΠ για να τη ζητήσουν να το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον εκτελεστικό κανονισμό. Επίσης, όσοι μετέχουν σε τέτοιες εκστρατείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ΠΕΠ αν έχουν ε, αρκετά μεγάλη πιθανότητα να επηρεάσουν την πολιτική. Μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει πάντα να προσπαθεί να αντιδρά στις επιτυχείς ΠΕΠ με συγκεκριμένες δράσεις και νομοθετικές προτάσεις. Επίσης και τώρα πάμε στο τεχνικό μέρος. Πολλοί πολίτες ε, φοβήθηκαν να υποστηρίξουν μια ΠΕΠ ε, διότι καλούνται να δώσουν αριθμό ταυτοτητήτων κλπ. Αυτό το είδαμε σε 18 χώρες. Ε, βλέπουμε ότι αυτή η ιδέα του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας δεν χρησιμοποιείται καν για να επαληθευτούν οι δηλώσεις υποστήριξη. Άρα δεν χρειάζεται στην πράξη. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό με τις 18 χώρες που τη ζητάνε. Ε, δύο λεπτά ακόμα, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ε, θα πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό του συστήματος συλλογής υπογραφών online. Ε, θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα και ο κύριος Πόλο θα μας τα πει αυτά σε ένα λεπτό. Επίσης οι θα πρέπει να συλλέγουν της ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποστηρικτών να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή δηλαδή με τους υποστηρικτές αυτό είναι σημαντικό και σημαντικό επίσης είναι να λαμβάνουμε υπόψη στα δεδομένα και τις απαιτήσεις προαπαιτούμενα ασφαλείας που υπάρχουν. πρέπει να επιλέγουν την ημερομηνία έναρξης μιας ΠΕΠ, θα πρέπει να μειωθεί η ηλικία για την υποστήριξη μιας ΠΕΠ στα 16, ε, Επίση θα πρέπει να δημιουργηθούν υπηρεσίε νομικέ, δηλαδή μια υποδομή που θα στηρίζει τις ΠΕΠ. Μεταφράσει, από την ΕΟΚΕ ευτυχώ μα είπαν ότι γίνονται, χρηματοδότηση ε, να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ε, μεταξύ πολιτών για τις ΠΕΠ. Πώς θα γίνει αυτό, με επιτυχημένες ΠΕΠ. Για να γίνει αυτό πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τον εφαρμοστικό κανονισμό της ΠΕΠ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και απαραίτητο νομικό καθεστώς για την ε, ευθύνη, για θέματα ευθύνης. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε νέα μορφή, να ανασχεδιάσουμε, να επανεκκινήσουμε την ΠΕΠ μπορεί έτσι να γίνει κινητήρια δύναμη για πιο συμμετοχική δουλειά σε, όλη, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή και θα δείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη, ότι οι ηγέτες της Ένωσης τους ακούν και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει θετικό ρόλο στη ζωή τους. Βλέπουμε ότι οι σημερινοί Ευρωπαίοι πολίτες δεν, δεν είναι ικανοποιημένοι αν ψηφίζουν κάθε πέντε χρόνια και μετά κάθονται στα παρασκήνια. Θέλουν να παρεμβαίνουν και ενδιαμέσω. Στο μεσοδιάστημα αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το παρατηρούμε μόνο εδώ στην Ευρώπη. Αλλά σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνηση, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, θέλουν οι πολίτε να παρεμβαίνουν και στο μεσοδιάστημα. Μεταξύ εκλογών ε, η μοίρα του, της ΠΕΠ είναι στα χέρια σας. Είστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι. Όπως είπε και ο κύριος Τίμαρμαν είστε η εθνική εταίροι. Ε, δουλεύετε εδώ και χρόνια για την εφαρμογή των ΠΕΠ και θέλουμε να σας ζητήσουμε να πάτε πέρα από τις περιορισμένες νομικές υποχρεώσεις που έχετε στα πλαίσια αυτού του επανελέγχου. Αναλάβετε πρωτοβουλία για θεμελιώδη μεταρρύθμιση και επανεκκίνηση της ΠΕΠ. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσει. Ε, γκρεμίστε τείχη που περιορίζουν τη συμμετοχική δημοκρασία, καταργήστε τους περιοριστικούς κανόνες ΠΕΠ και αφήστε να ακουστούν φρέσκες φωνές και ιδέες. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε πολλή ενέργεια ακόμα στην αίθουσα. Χαίρομαι. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέργκ. Ευχαριστούμε τη συνεισφορά σας. Τώρα με χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Φρανθίσκο Πόλο και εσείς 10 λεπτά έχετε. Καλημέρα σας. Είναι τιμή για μένα που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Δεθέρα που με επιτρέπει σήμερα να σας ε, παρουσιάσω τη δική μας ε, πρωτοβουλία. Θα συνεχίσω στα Ισπανικά. Στην πραγματικότητα δεν είμαι μόνος αλλά έχω μαζί μου 28 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που προσέτρεξαν στην πλατφόρμα μας τα τελευταία χρόνια για να εξωθηθούν αλλαγές. Και αν μάθαμε κάτι από αυτό είναι ότι οι πολίτες πραγματικά θέλουν να συμμετάσχουν και να συμμετέχουν. Προτού πάω στην ουσία της παρέμβασής μου θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα σχετικά με το τι συμβαίνει συνολικά στην πλατφόρμα μας. Το, Change είναι η μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα στον κόσμο. 85 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τη χρησιμοποιούν για να προωθήσουν αλλαγές που θέλουν να δουν. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα και ο καθένας μπορεί να επισημαίνει πράγματα που περισσότερο όταν ανησυχούν. Η Ευρώπη έχει σημαντικό ρόλο να διαματίσει το Change.org Περισσότεροι από 28 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι χρήστε σε χώρε όπω οι Ισπανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία. Η πλατφόρμα μα έχει ε, ε, τροποποιηθεί σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να ακούγεται η φωνή των πολιτών και να γίνονται, να προωθούνται οι αλλαγέ. Η χώρα λοιπόν από την οποία προέρχομαι και που ξεκινήσαμε στην Ευρώπη τουλάχιστον την change.org είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά χρηστών στον κόσμο της πλατφόρμας. Το 20% των χρηστών του ίντερνετ συνολικά στην Ισπανία είναι χρήστες του change.org. Σε όλες τις χώρες όμως οι χρήστες έχουν καταφέρει να τροποποιήσουν την νομοθεσία, να μπουν στην πολιτική ατζέντα και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό το έκαναν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία ε, πρωτοβουλία με πάνω από 300.000 υπογραφές ε, σχετικά με την ε, ευζοία των μελισσών και την καλύτερη διαχείριση του συστήματος. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις σημαντικότατες στοιχείες που, όχι, που δεν βρίσκουν πάντα την συνέχεια που θα έπρεπε να βρίσκουν στις επίσημες θεσμικές οδούς όπως οι πρωτοβουλίες. Καταρχάς, το ίντερνετ έχει άρρητα εμπόδια. Οποιοςδήποτε μπορεί να ηγηθεί μιας ε, πρωτοβουλίας για να αλλάξει κάτι. Και αυτό θα μπορούσε κανείς να το κάνει θέτοντας την πολιτική ατζέντα, τα τα θέματα που περισσότερο τον ενδιαφέρουν και τον ανησυχούν. Και αυτό ε, προκαλεί αλλαγές σε τέτοια ταχύτητα που βλέπουν οι πολίτες ότι η συμμετοχή τους πραγματικά αξίζει, αξίζει η προσπάθεια. Και θα ήθελα να εστιαστώ σε τρεις ε, βασικές ιδέες. Καταρχάς οι πολίτες συμμετέχουν όταν αυτό είναι εύκολο. Δεύτερον, συμμετέχουν όταν αυτό που κάνουν είναι χρήσιμο. Και τρίτον, θέλουν να γνωρίζουν οι πολίτες τι έχει γίνει μετά με τη συμμετοχή τους. Το πρώτο λοιπόν, η ευκολία της συμμετοχής σε, σε τρία μόλις χρόνια η change.org πέρασε από 10 εκατομμύρια χρήστες σε άνω των 85 και ο λόγος είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να παρέμβουν στην δημόσια συζήτηση, το δημόσιο διάλογο. Η ευκολία αυτή εξηγείται με τους εξής τρόπους. Καταρχάς η δημιουργία της αναφοράς, της αίτηση. Υπάρχουν πολύ απλά βήματα για μια εγγραφή αναφοράς και έχουν και συμβουλές και tips για να την κάνουν καλύτερα. Δεύτερον, είναι εύκολο να υποστηρίξει κανείς μια αναφορά, μια αίτηση, διότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης ταυτοποίησης και της ευκολίας των δεδομένων που ζητούνται όμως. Και τρίτον, είναι εύκολο να συμμετάσχει κανείς σε μια αναφορά, σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο όπως είναι ο δικός μας, ώστε να σωρεύεται στήριξη σε μια πρωτοβουλία. και ε, καμιά φορά υπάρχει μια υποτίμηση της ευκολίας του εύκολου τρόπου. Λες και το, όταν είναι κάτι εύκολο είναι λανθασμένο. Αλλά όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και περίπλοκα απομακρύνεται, απομακρύνονται οι πολίτες από την πολιτική διαδικασία. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτός. Πάω στο δεύτερο που είπα. Το χρήσιμο της συμμετοχής. Οι πολίτες μετέχουν όταν ξέρουν ότι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη διαδικασία, να τροποποιήσουν την κατεύθυνση. Η δυνατότητα ενός πολίτη να τροποποιήσει, να παρέμβει στην ε, νομοθετική διαδικασία περιορίζεται συνήθως από τους πολιτικούς μηχανισμούς, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες κοιτώντας σε πιο όριμες πρωτοβουλίες, προηγούμενες χρονικά πρωτοβουλίες όπως εκείνες που είχα, είχαμε στις ΗΠΑ, ε, πολύ συχνά ε, έχουμε όμως το φαινόμενο όπου έχουμε πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή. Στην Ισπανία υποβάλλονται πρωτοβουλίες από εκατοντάδες που έχουν υποβληθεί στην Ισπανία μόνο μία οδήγησε σε νομοθετική τροποποίηση. Στην change.org βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, την αντίθετη τάση. Οι χρήστες είναι εκεί για να προτείνουν νέα νομοθεσία και το επιτυγχάνουν. Άνω των 30 εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο έχουν συμμετάσχει με αναφορές που επέτυχαν να οδηγήσουν σε αλλαγές. Και με τις αλλαγές βλέπουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί δεν υπάρχει κανένα μεγαλύτερο κίνητρο για τη συμμετοχή από την επιτυχία, από το να ξέρει ότι αυτό που κάνεις οδηγεί σε αποτέλεσμα. Επίσης θέλουν να γνωρίζουν οι πολίτες τι έχει γίνει εκ των υστέρων με την υπογραφή τους, με τη συμμετοχή τους και θέλουν να το ξέρουν αυτό εγκαίρω. Μία από τις προκλήσει λοιπόν των ε, πρωτοβουλίων πολιτών είναι ακριβώς αυτή. Να γνωρίζουν οι πολίτες τι έχει συμβεί με τη συμμετοχή τους. Να γνωρίζουν πού κατέληξε αυτή η πρωτοβουλία και ότι δεν ήταν απλώ μία θεωρητική αναφορά ή ένα έγγραφο. Και ένας από τους βασικούς μηχανισμούς είναι η διευκόλυνση μέσω, μέσω επικοινωνίας άμεσης επικοινωνίας όλων των συνυπογραφόντων το οποίο αυξάνει το engagement λέει ο Μίλτης και ε, πλησιάζει περισσότερο στην πιθανότητα επιτυχία στην πρωτοβουλία το ίντερνετ μας προσφέρει όλα αυτά όλες αυτές τις δυνατότητες για να οδηγήσουμε σε αλλαγές, μια πλατφόρμα για την αλλαγή στην πραγματικότητα. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι πολιτικοί και οι θεσμοί μπορούν να ανταποκριθούν, μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα μηνύματα που τους δίνει το διαδίκτυο αυτή η ζωντανή κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ε, χρησιμοποιήσει ένα τεχνικό πλαίσιο ώστε να διαβιβάζονται όλα αυτά τα μηνύματα στους απαραίτητους πολιτικούς ηθήνοντες και να ακούνε τα μηνύματα των πολιτών. Και όλοι μπορούν να, γνωρί, να βλέπουν ζωντανά τι προσπαθούν να κάνει η ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή, σε άμεση επαφή με τους πολιτικούς ηθήνοντες, με αυτούς τους οποίους απευθύνουν το αίτημα την αναφορά τους. Η Κομισιόν δεν φαντάζομαι όμως ότι κάνει κάτι αντίστοιχο. Κάποιοι ευρωβουλευτές αυτής της αίθουσας, κάποιοι από τους ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου το κάνουν όμως ήδη μέσω της change.org. Εάν λοιπόν είδαμε κάτι σίγουρα σε όλες τις χώρες που, είμα, που έχουμε παρουσία είναι ότι όταν η πολιτική υποστηρίζει ε, τους πολίτες μάλλον όταν δεν δίνει απαντήσεις στις αιτήσει ε, των πολιτών, ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις οι πολίτες. Και τότε βλέπουμε μείωση των συμμετοχών στις ΕΠΕ, ε, στις ECI. Ενώ εμείς έχουμε τεράστια αύξηση. Δίνουμε έναν χώρο συμμετοχή στους πολιτών και γι' αυτό με μεγάλη χαρά θα συνεργαζόμασταν μαζί σας για να μπορέσουμε αυτή την πρωτοβουλία να την αποκαλέσουμε πρωτοβουλία των πολιτών ώστε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ένωσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τελευταία ομιλήτρια σε αυτό το πάνελ. Ε, πρωτού αρχίσουμε με τις ερωταπαντήσεις από τους συναδέλφους είναι η δόκτωρ Σουζάνα Ντελρίου Βίλιαρ. Σας δίνω τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Επιτροπή Βεβαίως Αναφορών. Το σύνολο της ε, ακαδημαϊκής μου δουλειάς από το διδακτορικό για τη συμμετοχή των ε, πολιτών, ε, της κοινωνίας των πολιτών μέχρι το σχέδιο το συνταγματικό της συνταγματικής συνθήκης σε όλη τη διαδρομή μου προσπάθησα να δώσω επιφάνεια στη σημασία της ε, συμμετοχής δημοκρατίας που συμπληρώνεται από την κοινοβουλευτική ή συμπληρώνει αν θέλετε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ ε, συνεργάζομαι με την Τροπία ΑΦΚΟ από πολλά χρόνια και μάλιστα σε μία από τις ε, συναντήσεις για τις πρωτοβουλίες πολιτών με τον κύριο Χάουρινγκ είχαμε μείνει εδώ είχαμε αποκλειστεί εδώ λόγω του εκείνου του ηφαιστείου στην Ισλανδία εν πάση περιπτώσει ε, θα ήθελα να πω ότι και ο κύριος Καζίνη και ο κύριος Γιολάινεν, ε, ο κύριος ε, Κάστεμπεργκ πάρα πολλοί ευρωβουλευτές πάρα πολλοί συμμετέχοντες από τον ακαδημαϊκό χώρο έχουν δουλέψει, έχουν εργαστεί ώστε να βρίσκεται εδώ η πρωτοβουλία των πολιτών. Τώρα, γιατί πιστεύω στο πρόγραμμα αυτό Upgrading Europe, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται μια αναβάθμιση επιφάνειας ή στα μάτια των πολιτών. Και πραγματικά διεθνική, υπερκρατική, οριζόντια δημοκρατία είναι μια δημοκρατία πολύ ισχυρή. Και με την συνθήκη της Λισαβόνας ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε την επιρροή του και επομένως ενισχύθηκε και η επιρροή των πολιτών μέσω αυτού. Και εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά στο 47-7 ότι ε, συμπεριελήφθη το πέρασμα για την συμμετοχική δημοκρατία, όπως και για την νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών που τότε απεκλήθη με αυτό το όνομα. Και είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται η λέξη νομοθετική, γιατί έτσι καλείται η Κομισιόν να εκκινήσει μια νομοθετική διαδικασία. Το 47 άρθρο λοιπόν το οποίο αφιερώνεται στην συμμετοχική δημοκρατία που συμπληρώνει το 46 την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στον τίτλο 4 ήταν σίγουρα μία από τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν επιτυχίες. Αλλά πέρα από τεχνικά και νομικά ζητήματα από τα οποία έχουμε μάθει πολλά και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι οι ακαδημαϊκοί και βουλευτές πέρα από όλα αυτά τα θέματα πρέπει να εστιαστούμε στην ίδια τη διαδικασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών από το 2002 μέχρι το 2012 1η Απριλίου όπου εκείνη η πρωτοβουλία είναι μια διαδικασία πραγματικά αξιολογότατη Γι' αυτό το λέω ε, το έχω γράψει και στο καινούργιο μου βιβλίο που στις 15 Ιανουαρίου παρουσίασε εδώ στο Κοινοβουλίο και που ε, οπωσδήποτε ε, περιγράφει την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών η οποία ΠΕΠ ECI πρέπει να είναι σαφής και να είναι κάπως πιο εύκολη στη χρήση της το θέμα της συλλογής των υπογραφών, των, ε, της επικύρωσής τους κτλ. είναι σημαντικό, αλλά η πρωτοβουλία των, των Ευρωπαίων πολιτών δημιουργεί μια δυνατότητα πολύ σημαντική διότι ανακαλεί το λόγο για τον οποίο ε, δημιουργήθηκε. Η ισχύ λοιπόν που έχει η ECI είναι ισχύς ως προς την επικοινωνία ως προς την επικοινωνία και τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Αυτό λοιπόν θα ήθελα κυρίως να τονίσω προς το ακριατήριό μου σήμερα. Οι πολίτες συμμετέχουν με ένα κεντρικό τρόπο ε, και συνθετικό τρόπο και έχουν τόσο μεγάλη ε, επικοινωνιακή ισχύ αυτές οι πρωτοβουλίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα θεσμικά όργανα τις πρωτοβουλίες αυτές ώστε να επικοινωνήσουν καλύτερα και πιο άμεσα με τους πολίτες. Και γιατί το λέω αυτό, διότι η πρωτοβουλία με αυτή την συλλογή υπογραφών ενός εκατομμυρίου σημαντικών αριθμών δηλαδή πολιτών και εγώ θυμάμαι πολύ καλά όλες τις ε, συνεδριάσεις σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να είναι αυτός ο σημαντικός αριθμός και ποιος ο απαραίτητος αριθμός των χωρών που θα έπρεπε να συμμετέχουν σε πρωτοβουλία ώστε να μπορεί να θεωρείται υπερεθνική πρωτοβουλία πολιτών όλα αυτά έχουν την εξής δύναμη ώστε η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών να έχει ένα πραγματικό πράσινο φως και ώστε η Κομισιόν να μπορεί να την εγκρίνει οι πολίτες που υπογράφουν την ε, ECI και οι διοργανωτές της θα πρέπει να ενημερωθούν και ταυτόχρονα να ενημερώσουν σχετικά με τις κεντρικές αξίες Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία τη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με ένα θέμα στο οποίο έχω εστιαστεί τελευταία, σχετικά, για παράδειγμα, με την αναθεώρηση των πρωτοβουλειών αυτών, οι οποίες δεν ανακρίθησαν τελικά. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να πω ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι εκείνες οι πρωτοβουλίες που δεν κατάφεραν να πάρουν το πράσινο φως για τεχνικούς λόγους συλλογής υπογραφών, χρονισμού, πρόσβασης ή οτιδήποτε άλλο, είναι αλήθεια ότι ίσως θα έπρεπε να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Όμως στη δημοκρατία δεν είναι ότι ισχύουν τα πάντα, ότι όλα είναι καλά. Και μάλιστα τελευταία έχουμε ανησυχητικά σημάδια για τη δημοκρατική πορεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως όλα αυτά τα φίλτρα που έχουν σχέση με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, με τη λειτουργία και με τον τρόπο λήψης αποφάσεως από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του διαλόγου για το πώς πρέπει να κάνουμε υπερ πολιτική Όλα αυτά πρέπει να διατηρούνται, διότι στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες, δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι θέλουμε. Επανέρχομαι λοιπόν στην ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία που συμπληρώνεται όπως έλεγα από, τον, ε, από τη συμμετοχή εκεί. Ακριβώς αυτό ήταν το θέμα του διδακτορικού μου που σας έλεγα και, ε, και πολλών από τις δημοσίευσεις μου όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να ηγηθεί η συμμετοχή, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, διότι πρέπει να ανακτηθεί ε, έδαφος σχετικά με το τι πρέπει να σημαίνει η δημοκρατία, ποιες είναι οι προκλήσεις που είναι πάρα πολλές και πολύ σημαντικές σε αυτά που αντιμετωπίζουμε η Ευρώπη των πολιτών, η Ευρώπη η πρακτική, η Ευρώπη η χρήσιμη είναι βεβαίως πολύ σημαντικά και επομένως μία πλατφόρμα, ένας νέος οδηγός σχετικά με το πώς πήγαν τα πράγματα αυτά τα χρόνια, τι επιτύχαμε, τι όχι, ποια υπήρξε η διαδικασία της γέννησης αυτής της, ε, του θεσμού της πρωτοβουλίας των ε, Ευρωπαίων πολιτών με εκπροσώπους οργανώσεων, μη κυβερνητικών φορέων κτλ είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα βήμα, ένα φόρουμ, μία πλατφόρμα στο οποίο να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι οι προκλήσεις, τι είναι αυτά που πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν ώστε να συνεχίσει να υφίσταται ένα μέσο, ένα εργαλείο τόσο πολύ σημαντικό. Και επαναλαμβάνω το εξής Η ισχύση επικοινωνιακή που έχει η πρωτοβουλία των πολιτών η ισχύση νομοθετική ώστε να, προταθούν συγκεκριμένες να αναλυφθούν μάλλον συγκεκριμένες νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες και προτάσεις και βεβαίως κοινοβουλευτική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία που θα συμπληρώνεται από τη συμμετοχική δημοκρατία. Και ο William Butler Gates όπου τότε ήταν πρόεδρος ο Πατ Κόξο και αναφέρθηκε στο Γέιτς. όπου είπε προχώρησε προσεκτικά γιατί, προ, γιατί πατάς βηματίζεις πάνω στα όνειρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah, we must all thread... Πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σχετικά με την βελτίωση αυτού του εργαλείου. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και για το στοιχείο που αναφέρατε της συμμετοχικής δημοκρατίας που πρέπει να το τονίζουμε ε, συνεχώς. Σας ευχαριστώ και τους τρεις για τις παρεμβάσεις σας που ήταν πάρα πολύ χρήσιμο που σας ακούσαμε. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω παρεμβάσεις από τα μέλη των επιτροπών και από άλλες επιτροπές που μπορεί να είναι εδώ για ερωτήσεις. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Γκέραρτ. Χαίρομαι που χαιρετίζω ε, και πάλι τον κύριο Χέφνερ, ο οποίος ήταν από τα βασικά μέλη όταν αυτό εκπονήθηκε η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και εκ μέρου των Πρασίνων που θέλανε πρόσθετο χρόνο. Σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Σεσίλια, Ντανούτα και για όλους. Για... Θα ήθελα να θέσω ένα απλό ερώτημα. Όταν μιλάμε ε, για την εξακρίβωση των υπογραφών, πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πολίτες που θέλουν να υπογράψουν. Πρέπει να ξέρουν τι χρειάζεται για να υπογράψουν. Όταν εκπονήσαμε τον κανονισμό θέλαμε ένα, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για όλη την Ευρώπη με ονόματα ε, διεύθυνση και υπογραφή και μου είπανε ότι δύο κράτη-μέλη δεν μπορούν να το δεχτούν. Εκείνη την εποχή είπαμε εντάξει, ας κάνουμε μια εξαίρεση για αυτούς που απαιτούν διαφορετικά στοιχεία, αλλά μέσα σε τρία χρόνια θα έπρεπε να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο και να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για την πρωτοβουλία. Και θα ήθελα να μάθω τι συνέβη εντωμεταξύ και δεν πέτυχε αυτό. Τι κάναν αυτές οι χώρες, τι έκανε το Συμβούλιο, τις Επιτροπές, ώστε να είναι φιλική προς τους πολίτες αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση. Ο κύριος Τεραμπράς έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. ε πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία ε, και η έλλειψη υποστήριξης ε, νομικής ε, και διοικητικής μέρημνας παρεμποδίζει τους Ευρωπαίους πολίτες. Υποστηρίζουμε πλήρως τις 10 συστάσεις του κυρίου Μπέργκ, χωρίς κανένα περιορισμό, καμία επιφύλαξη. Αυτές οι 10 και άλλες παρόμοιες συστάσεις δεν θα έχουν ως άμεση επίπτωση όλα οι πρωτοβουλίες να επιτυγχάνουν. Ούτε και καμία ίσως, αλλά πάντως αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός πραγματικού πλέγματος ε, ενέστησης ε, και ε, συμμετοχής μεταξύ ε, των πολιτών. Ε, η πολιτική είναι παιδαγωγική, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ και εγώ. Καταρχήν μια ερώτηση. Και το γεγονός της διοργάνωσης αυτής της ακρόασης από μόνο του δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι βουλευτές θεωρούν πολύτιμη την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και τη θέλουν και στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντική προσθήκη ενός δημοκρατικού κράτους ότι μπορούν άμεσα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι πολίτες. Επίσης, κάθε τυπικό εμπόδιο πρέπει να εξαλείφεται γιατί βέβαια ε, ε, έχουμε 28 ε, τροπολογίες για να βελτιωθεί ή να πλουστευτεί ο κανονισμός. Όλες οι πρωτοβουλίες που δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες υπογραφές θα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία μιας συνήθους αναφοράς. Ενδεχομένως αυτό να είναι μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ, κύριος Γιώχανσον. Οι περισσότερες διαδικασίες ή τουλάχιστον ένα μέρος τους θα κατέπιπταν αν στον κανονισμό και στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διατύπωση εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούσε να αντικατασταθεί αυτή η διατύπωση όπως πρότεινε και ο Γιώ Λάινεν με το εκτός αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών συνθήκων. θα περίτευαν πολλές διαδικασίες και προσφυγές στο δικαστήριο, αν γινόταν αυτό. Προτείνω να σκεφτούν οι δύο επιτροπές αυτό το ενδεχόμενο, να κάνουν πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, αυτή την τροποποίηση στην ε, συνθήκη. Σχέδιο τροποποίηση στη συνθήκη δηλαδή. Η κυρία Μέρτς. Να απαντήσω στην ε, πρόταση πρωτοβουλίες που απέτυχαν, όπως λέγονται, μπορούν να γίνουν αναφορές. Η πράξη θα δείξει την επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Υποθέτω εκ πείρας ότι είναι σημαντικό να πούμε στους υπογράψαντες ότι δεν χάθηκε η προσπάθειά σας. Κομισιόν μπορεί να μην ανέλαβε δράση, αλλά το πρόβλημά σας θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω δηλαδή ότι έτσι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Ο κύριος Χαουριέγκο. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τους εμπειρογνώμονες βλέπουν δυνατότητα ε, όχι όλες οι ΠΕΠ να οδηγήσουν σε νέο, νέα νομοθεσία αλλά αν ανοίξει αυτή η διαδικασία και αν απαλληφθούν πολλά εμπόδια και φίλτρα μπορεί οι προτάσεις που προέρχονται από τους πολίτες όχι όλες αλλά πολλές από αυτές να μπορούν να μετατρέπονται σε νομοθεσία ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες ε, που ήρθαν να μας βοηθήσουν και τους ρωτώ αν θεωρούν ότι ε, θα μπορούσαν πολλές από τις εύλογες προτάσεις να ακολουθήσουν άλλες διαδικασίες όπως στάσεις προς κυβερνήσεις. Ένα παράδειγμα. Οι άλλες οδούς, γιατί αν δεν γίνει αυτό δεν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία. Δηλαδή αρχίζει μια διαδικασία, μετά μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα αρμοδιότητας και μπορεί ε, για λόγους επικουρικότητας πολλές φορές ε, και σχετικών εμποδίων να σταματάει η διαδικασία. Πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες ότι υπάρχουν άλλες εναλλακτικές Μπορεί δηλαδή να μετατραπούν όχι μόνο σε νόμο οι πρωτοβουλίες αλλά και άλλα πολιτικά μέσα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο κύριος Γέρι Βάιερ, αν είναι μαζί μας. Ναι, ευχαριστώ. Σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό. Εγώ είμαι σε εκστρατείας Είμαι από το Λουξεμβούργο και είμαι στους δρόμους στο Λουξεμβούργο ε, και κάνω εκστρατεία για διάφορες πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών. Προτού εξηγήσω ποιος είναι ο σκοπός μια συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, πρέπει πρώτον να εξηγήσω τι είναι η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα προώθησης του μηχανισμού αυτού που δεν είναι γνωστός από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες που έχουν δικαίωμα να υπογράψουν ή ε, να λανσάρουν μια πρωτοβουλία. Οι δυνατότητες λοιπόν συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών είναι σημείο το οποίο θα πρέπει ε, να τονιστεί και να διευθυνιστεί στην έκθεση όταν μιλάμε για την πρωτοβουλία. Ότι όλα αυτά δεν έγιναν με τρόπο που συνάδει με τον στόχο της προώθησης της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών. Μ' αρέσει η ιδέα του καθηγητή Σωρό να έχουμε ένα ε, σημείο στην ημερήσια διάταξη των Συμβουλίου για το θέμα αυτό, να οργανώσουμε τοπικές συναντήσεις, τοπικές ε, εκστρατείες για να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, να υπάρχει μια, μια βάση δεδομένων ε, για επικοινωνία, για να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, για υποστήριξη. Θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το μηχανισμό αυτό. Ε, είμαστε πολιτικοί και όλοι πρέπει να πάρουν στα σοβαρά την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών για να δείξουν πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες μας και τα συμφέροντά τους. Σας ευχαριστώ ε, για τις, ε, τη συμβολή σας. Α, Σαρτ Γκέρενς, σας δίνω το λόγο. Ναι, απαντώ μια σκέψη που έγινε σχετικά με την δυνατότητα παρα, ε, παρα, παραδοχής μιας αίτησης. Γιατί να μην δεσμευτούμε το αίτημα να υποβάλλεται εκεί όπου είναι αρμόδιο το όργανο, ούτω ώστε οι πολίτες να εισακούονται αν έχουν ένα πρόβλημα. Ε, βεβαίως ε, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται αν είναι το τοπικό επίπεδο, το εθνικό ή το ευρωπαϊκό. Ε, όποιος μπορεί να έχει αρμοδιότητα στον τομέα αυτό θα πρέπει να απαντήσει και αυτό γίνεται σε όλες τις εθνικές δικήσεις αν στείλετε κάτι σε ένα διοικητικό όργανο που δεν είναι αρμόδιο έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει το αίτημα αυτό στο αρμόδιο διοικητικό όργανο να το πράξουμε αυτό ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει την εντύπωση ότι δεν λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ και τώρα ε, δίνω τον λόγο στην κυρία Αλτά. Ναι, παρακολούθησα όλη τη συζήτηση το πρωί και νομίζω ότι κάτι δεν είναι σαφές για μένα ένα από τα προβλήματα της πρωτοβουλίας ότι παρουσιάζεται ε, πολύ συχνά στους πολίτες ως μέσο επιρροής. Δεν είναι σωστό αυτό. Και ενώ δεν λέμε, λέμε ε, ότι αν δεν αποφασίσει ένα εκατομμύριο τι συμβαίνει. Αλλά ενώ λέμε στους ανθρώπους μιλάμε με αυτή τη γλώσσα ότι μπορούν να έχουν επιρροή, βεβαίως στο τέλος θα αισθανθούν απογοητευμένοι. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί για τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Δεύτερο σημείο, ένας λόγος για την έλλειψη εμπιστοσύνης της δημοκρατίας μας είναι η διαφθορά. Είναι η ε, φοροδιαφυγή είναι ε, το η έλλειψη διαφάνειας κλπ. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά ε, να, με το, με αν θα μπορούμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία των δημοκρατιών μας, όχι, δεν νομίζω. Και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Κέρτον Ντόλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω δεν αισθάνομαι καλά με την ε, ιδέα του να βάλουμε στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην μερίσια διάταξη. Αλλά μια φορά το χρόνο να ακούμε τους πολίτες ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να μην τους ακούμε συνεχώς. Το μήνυμα αυτό είναι περίεργο. Το άλλο θέμα είναι που πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη για τις τεχνικές προοπτικές είναι ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων διότι κυρίως αν σκεφτούμε τα όσα αλλάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτοί οι μεγάλες οργανώσεις εκστρατιών στο διαδίκτυο πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα από το πώς συμπεριφέρονται και εμείς τα ευρωπαϊκά όργανα έχουμε εξουσία στα χέρια μας, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο οπαδούς στα κοινωνικά δίκτυα δεν λέω για διαφήμιση, αλλά θα μπορούσαμε να διαδώσουμε πολύ περισσότερο την ιδέα αυτή, μια εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα των σκέψεών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους ε, εμπειρογνώμονες για ένα λεπτό καθένας για συμπεράσματα. Ο κύριος Μπέργκ πρώτα απ' όλα. Κάρστεν Πρώτο θέμα. Βεβαίως όλες οι πρωτοβουλίες δεν οδηγούν σε νομοθετικές ε, προτάσεις. Είναι φυσικό, αλλά καμία πρωτοβουλία δεν οδήγησε ε, σε πρόταση. Η συνέπεια λοιπόν είναι μία αλλαγή, έλλειψη αλλαγής. Θα πρέπει την αντίληψη του, ε, της ΠΕΠ ε, να την λάβουμε υπόψη σοβαρά και να αρχίσει η νομοθετική διαδικασία από την Επιτροπή, τουλάχιστον να το βάλουμε στην ατζέντα ε, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μόνο τότε ε, θα είναι το θέμα ελκυστικό για τους πολίτες. δελειώς τα πράγματα δεν είναι σοβαρά σχετικά με την ερώτηση Χέφνερ. Μιλάμε τώρα για τεχνικά πράγματα. Ξέρετε ότι το παράρτημα 3 του κανονισμού λέει ότι μπορούν να αλλάξουν οι προϋποθέσεις από τα κράτη και είναι υποχρεωμένες να το πράξουν αν δεν συνάδουν με τις υπόλοιπες. Ε, ε, το Λουξεμβούργο ε, μείωσε το, το, το περιορισμούς, θα πρέπει και οι άλλες χώρες να κάνουν το μάθημά τους, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. να απαντήσω στην παρέμβαση του κυρίου Χάργκλης. Αν θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τις πρωτοβουλίες που δεν λειτουργούν σε κάτι άλλο. Η απάντησή μου είναι όχι, όχι και ακόμα όχι. Οι πολίτες θέλουν να δουν πραγματικές αλλαγές. Ενδιαφέρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν ενδιαφέρονται για, για τα τεχνικά εμπόδια ή την αρχή της επικουρικότητας ή τα προβλήματα που έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς εδώ. Τους ενδιαφέρει να βελτιώσουν τη ζωή τους. Εάν οι θεσμοί δεν είναι οι κατάλληλε δίωδοι για να τροφοδοτηθεί η αλλαγή αυτή, θα δούμε αυτό που ακριβώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ότι θα διοχετευτεί αυτή η προσπάθεια σε άλλες διόδους, σε άλλα κανάλια. Θα εκστρατεύσουν και θα διαδηλώσουν έξω από τα σπίτια ίσως των ε, πολιτικών εθνών και των βουλευτών. Θέλουν πραγματική αλλαγή οι πολίτες. Η κυρία Βιγιάρ έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, τα εξή δύο. Καταρχά για το, για το θέμα της ε, επικοινωνίας. Πράγματι έχουν πολύ ε, σημαντική δυναμική οι πρωτοβουλίες υπό την έννοια αυτή και βεβαίως θα πρέπει να επικοινωνούμε πολύ περισσότερο με τους πολίτες ώστε να ενημερώνουμε μέσω τηλεοράσεων, ραδιοφώνων κτλ. σε τι συνίσταται η πρωτοβουλία των ευρωμένων πολιτών. Και για την ε, πολύ σημαντική πρόταση σχόλιο του ε, ε, Ραμόν, ναι θα έλεγα υπάρχουν πρωτοβουλίες που ίσως κάποια στιγμή δεν εγκρίνονται για μια σειρά από παραμέτρους της Κομισιόν μεταξύ άλλων, αλλά το να μην μένουμε σε ένα συγκεκριμένο στενό πλαίσιο και συγχρονισμό μεταξύ των διατάξεων των εθνικών και των ευρωπαϊκών κανονισμών, ακόμα και αν ισχύουν όλα αυτά, πρέπει να εξακολουθούν να έχουν επιφάνεια οι προσπάθειες αυτές, οι πρωτοβουλίες αυτές. Η κυρία Γουάλης που κάθεται δίπλα μου, ο κύριος Καζίνη, οι ευρωβουλευτές το γνωρίζουν πολύ καλά στην ανάπτυξη ε, του χάρτη, της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων για παράδειγμα όπως και της ε, συνταγματικής συνθήκης ακούστηκαν πάρα, πολύ πολλές ιδέες που σε κάποια, σε, σε κάποια χρονικά παρεάσματα της νίκης για παράδειγμα δεν ήταν δεσμευτικά ενώ ακολούθως η Νικόλ Φοντέν είπε ότι η χάρτα Θεμελιωδών δικαιωμάτων θα ήταν το φύλλο πορείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή τη στιγμή η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι νομικά δεσμευτική και προσαρτημένη στην συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω να πω ότι πολλέ ιδέε και πολλέ προτάσει, που υποβάλλουν οι πολίτε ίσω σε μια πρώτη χρονική στιγμή μπορεί να μην εγγράφονται, μετεγγράφονται σε μια νομική διάταξη, σε μια νομοθετική διάταξη, αλλά εγώ από τις εργασίες μου τις ακαδημαϊκές γνωρίζω ότι αργότερα ίσως σε μια δεύτερη φάση αυτές οι ιδέες πράγματι μπορούν να ενσωματωθούν και να μετεγγραφούν στις, ε, στους κανονισμούς μας, στη συνθήκη μας και λειτουργούμε υπό αυτές τις νομικές διατάξεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με αυτό ολοκληρώνεται το πάνελ αυτό. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Ήταν εμπνευσμένα όλα αυτά που ακούσαμε και ξαναδίνω το λόγο στην Τανούτα για να μας εισαγάγει τα μέλη που εργάζονται και τα τωρινά και τα του παρελθόντος. Ευχαριστώ πολύ. Σε, αυτό το, σε αυτή τη συνεδρία έχουμε πραγματίσει συγητές παλιούς και νυν η πρώτη η ομιλήτρια είναι η κυρία Νταϊάννα Βόλις. Παρακαλώ να τηρήσουμε τα χρονικά περιθώρια. Ευχαριστώ, θα κάνω το καλύτερο. Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε πάλι εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Ήταν από τις κορυφαίες στιγμές της σταδιοδρομίας μου η συμμετοχή μου στη συγγήτρια στο ΠΕΠ μην ξεχνάμε και την εποχή... Ε, ε, μην ξεχνάτε και ότι επιλέξαμε τέσσερις εισηγητές να έχουμε από, τις, από δύο πολιτικές ομάδες. Ε, αυτό απέδειξε τη σημασία που αποδίδαμε στο θέμα και βεβαίως το μήνυμα που θέλαμε να αποστείλουμε. Και τότε και τώρα ήμουν ένθερμη θειασότης της διαδικασίας αυτής. Είχαμε μια ευκαιρία για συμμετοχική δημοκρατία, είχαμε μια ευκαιρία να πούμε στους πολίτες ότι δεν ε, έχετε μόνο τη δυνατότητα να ε, κάνετε καταγγελίες αλλά να πατήσετε και το κουμπί της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό ήταν κεντρικό στο μυαλό μας σχετικά με το τι θέλαμε να πετύχουμε. Πριν έρθω εδώ σήμερα σκεφτόμουν την εμπειρία μου, τις παρατηρήσεις που ε, έκανα τον τελευταίο καιρό εκτός Κοινοβουλίου. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι υπέγραψα online μια πρωτοβουλία πολιτών. Δεν θυμάμαι ακόμα και τώρα και ακόμα και σήμερα ποια ήταν, γιατί δεν είχα ανάδραση, δεν υπήρξε διάλογος και αρχικά είχα σκεφτεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει συμμετοχή, να υπάρχει διάλογος, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έτσι λοιπόν, εκεί που καθόμουν σπίτι μου και έπινα τον καφέ μου, σκεφτόμουν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, Ενδεχομένω είναι πιο εύκολο εγώ να απευθύνω επιστολή στον, σε έναν επίτροπο ή στον διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο ή σε ένα μέλος του Κοινοβουλίου. Γιατί να αρχίσω μια πρωτοβουλία πολιτών. Όμως σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία έλεγα ξανά και ξανά πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία για την επαφή μας με τους πολίτες. Οπότε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είπαμε πολλές φορές σήμερα ότι ε, θα πρέπει ε, ε, όπως λέει και το προήμιο να είναι απλές, σαφείς, φιλικές προς τον χρήστη και τον πολίτη. όπως είπε και ο Ζέραλ Χάφνερ, είπαμε ότι θέλαμε κάτι που να είναι το ίδιο σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλαμε τις υπογραφές να τις αποφασίζουν οι πολίτες πώς θα γίνει τη διαδικασία, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα απλό σύστημα. Αυτό είναι το ζητούμενο για να έχουμε ευρωπαϊκό μέσο σαφές, σαφές και φιλικό προς τον χρήστη. Αυτός ήταν αρχικά ο σκοπός μας και αυτό πρέπει να επιτύχουμε. Βεβαίως δεν θέλω να θεωρήσετε ότι είμαι απεσιόδοξη αφού πιστεύω ότι η δυναμική υπάρχει στο μέσο αυτό ακόμα για να εξασφαλίσει και να προωθήσει το διάλογο σε όλες τις ε, περιπτώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά υποπτεύομαι, αν σκεφτώ και το δικό μου το κράτος μέλος, στη δική μου τη χώρα, ε, δεν ε, έχουμε συνηθίσει να μας λένε ότι έχουμε το δικαίωμα να ε, ε παίρνουμε πρωτοβουλίες για νομοθεσίες. Ε, έχω δει πολλές αναφορές για ένα σωρό παράδοξα πράγματα, αλλά η ιδέα ότι μπορούμε να ε, δώσουμε ένα κτίριο λάκτισμα για να ε, υπάρξει νομοθεσία, αυτό σημαίνει μεγάλη ενημέρωση. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε για αυτήν και ενδεχομένως μετά να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ Νταϊάννα και τώρα ο Κάρλο Καζίνη, πρώην πρόεδρος της, Ευρωπα... της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. Συγγνώμη Κάρλο, μόνο πέντε λεπτά μπορώ να σου δώσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ όχι μόνος πρώην πρόεδρο ε, της Επιτροπής παρεμβαίνω, αλλά και βεβαίως η Επιτροπή έχει δουλέψει πολύ στον κανονισμό 2.11, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλα τα θεσμικά όργανα, με άλλους θεσμικούς προσώπους, όπως και με την συνέλευση των Εθνικών Κοινοβουλίων, την ΚΟΣΑΚ. Αλλά θα ήθελα να τοποθετηθώ ιδιαίτερα σε σχέση με την πρωτοβουλία One of Us. διότι είναι αν θέλετε το παράδειγμα των όσων πρέπει να αλλάξουν αυτή η πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία συνέλεξε πάνω από 2 εκατομμύρια υπογραφές, δηλαδή περισσότερο από όλες τις άλλες πρωτοβουλίες των πολιτών. Άκουσα από την Κομισιόν τους αριθμούς 50, 26, 26 δηλαδή που κατεγράφησαν ε, και δύο που υπερέβησαν τελικά το, το τελικό φίλτρο εξέτασης. Η Us, λοιπόν σε 19 χώρες ε, ξεπέρασε το ελάχιστο όριο του κανονισμού άνω των 2 εκατομμυρίων και τελικά επικυρώθηκαν 1 εκατομμύριο 890 τόσες χιλιάδες. Μόνο στην Ιταλία είχαμε 150.000 ε, υπογραφές που δεν τη διαβίβασε διότι δεν υπήρχε η κατάλληλη αδειοδότηση ο Ιταλικός φορέας. Δηλαδή και αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Εγώ δεν είμαι υπέρ των, της μείωσης των ελέγχων εγκυρότητος ή σοβαρότητος, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται πράγματι για μια πραγματική προσπάθεια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάτι να κάνουμε και διαβάζοντας ε, τον κανονισμό 2.11 και την συνθήκη Λισαβόνας είναι, όλα είναι σαφέστατα. Θα πρέπει να πλησιάσουμε στους πολίτες για να έχουν, και διαβάζω πραγματικά το προήμιο του κανονισμού, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να ε, δημιουργηθεί μια συνείδηση πολιτική ευρωπαϊκή. Αλλά η επίπτωση της πορείας της One of Us ήταν ακριβώς η αντίθετη. Ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνη, η καχυποψία διότι είδαν ότι οι προσπάθειές τους πήγαν χαμένες. Ήταν ένα ρήγμα δημοκρατικό, διότι ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων ματέωσε την προσπάθεια άνω 2 εκατομμυρίων, ε, χωρίς να γίνει και κάποιος διάλογο στη συζήτηση. Ο κίνδυνο λοιπόν είναι όχι μόνο δεν θα πλησιάσουμε του πολίτε, αλλά το αντίθετο θα γίνει. Και το σφάλμα είναι στο, στο 10 σε του κανονισμού και υποβάλλω συγκεκριμένε προτάσεις. Το στοιχείο σε λοιπόν δίνει το δικαίωμα στην Κομισιόν να αναλάβει δράση ή όχι. Οι πολίτες περιμένουν όμως ότι τα θεσμικά όργανα, μεταξύ των οποίων και το Κοινοβουλίο, να απαντήσει στις προσδοκίες τους. Και εδώ έχουμε κριτήρια παραδεκτού της Κομισιόν προκειμένου να αποδεχθεί όχι μια, μια τέτοια αίτηση, μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά οι λόγοι για τους οποίους η Κομισιόν έλεγε τελικές ανακοινώσεις ήταν οι ίδιες που ήταν στην αρχή. Μπορούσαν να καταχωρήσουν. Γιατί τελικά λοιπόν να καταβάλει κανείς όλη αυτή την προσπάθεια αν είναι να ματαιωθούν τα πάντα. Ο κανονισμός προβλέπει ένα πεδίο περιορισμού των καταχωρήσεων που θα μπορούσε και να, να απλουστευτεί λίγο. Αλλά πάνω από όλα εδώ πρέπει να σκεφτόμαστε το εξή η πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Ε, κάτι σαν δημοψήφισμα, λαϊκό δημοψήφισμα, το οποίο έχει κριτήριο παραδεκτού, αλλά έχει και υποχρεωτική επιρροή νομική, επίπτωση. Ενώ στην αναφορά στην πρωτοβουλία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έλεγχο και ε, ω εκ τούτου μπορεί και να την αγνοεί κανεί ολοκληρωτικά. Αλλά δείτε και τις αναφορές που έχουμε στο Κοινοβουλίο. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να πλησιάσουμε τις πρωτοβουλίες, τις αναφορές, τροποποιώντας το άρθρο 10 και ίσως και το 11 του κανονισμού. Επί της ουσίας χρειάζεται υποχρεωτικότητα σημαντικού, σημαντικής συζήτησης, ευρεία συζήτησης στο Κοινοβουλίο και ίσως και στα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο άρθρο 11 της συνθήκης γίνεται επίκληση στην Κομισιόν να υποβάλει. Αλλά πρόκειται για πρόσκληση, πρόσκληση στην Κομισιόν. Δεν έχουμε συνέπειες δηλαδή για μη υποβολή τέτοια από Κομισιόν. Εκφράζει η Κομισιόν της θέσης ε, της ή μια γνωμοδότηση ή μια ανακοίνωση ή οτιδήποτε άλλο δεν διαφημίζει η συνθήκη της Λισαβόνας τι νομικό μέσο πρέπει να είναι, αλλά πρέπει να το κάνει. Επομένως χρειάζεται μια, ε, ένας διάλογος κοινοβουλευτικός και πρέπει να δούμε επίσης πιο συγκεκριμένα ποια είναι η διαφορά της ε, πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών που υπογράφει άνω του ενός εκατομμυρίου κτλ. και της αναφοράς. Αναφορά μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, χωρίς να υπάρχει νομική δεσμευτικότητα και εφόσον υποβληθεί από του πολίτε, πρέπει να συζητηθεί ή στο κοινοβούλιο. Επομένω, αυτέ οι διαφορέ πρέπει να τονιστούν, πρέπει να εξεταστούν. Και ζητώ τελικά και ω πρώην πρόεδρο και ω εμπειρογνώμονε σε αυτά τα θέματα να σκεφτούμε πολύ σοβαρά του, την τροποποίηση του 10 και 11 του κανονισμού 2.11. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Κάρλος. και καταλαβαίνω ότι και οι τωρινοί εισηγητές σας άκουσαν με προσοχή δίνω τον λόγο στον Γιώργη Τσόπφλιν που είναι εισηγητής για την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βρίσκω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, πολύ πλούσια σε γνώσεις, έμαθα πολλά ε, σημείωσα με προσοχή πολλά από τα οποία λέχθηκαν και θα τα περιλάβω στην έκθεσή μου. Αλλά το σημείο κίνησης είναι μια ρητορική ερώτηση αν θέλετε. Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτυχία. Όχι δεν είναι αποτυχία αλλά δεν είναι και επιτυχία. Διότι αν ήταν αποτυχία θα έπρεπε να την παραμερίσουμε. Είναι λοιπόν ένα σημείο κίνησης και θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε. Και αυτό, αυτές είναι οι σκέψεις που θέλω να σας προσφέρω, πρακτικές και άλλες. Έχω την, ε, την εντύπωση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο ειδικό σε κάθε κράτος μέλος για να βοηθάει τους πολίτες για να υποβάλουν, για να οργανώσουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Κυρίως τα μεγάλα κράτη. Ε, βεβαίως, ε, εμεί οι Ούγγροι είμαστε ανάμεσα στα μεγάλα και στα μικρά κράτη. Πρέπει να υπάρχουν τεχνικές συμβουλές ε, για αυτούς ε, που σκέφτονται να οργανώσουν μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Ποιες είναι οι παγίδες, ε, ποια είναι τα εμπόδια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση που σταματάει η πολιτική, το πολιτικό τομέα και που αρχίζει ο νομικός, ο τεχνικός. Υπάρχει ένα πρόβλημα που υπάρχουν νομικά θέματα, που υπάρχουν πολιτικά θέματα και υπάρχει το μείγμα των δύο έχει προκαλέσει τόσες πολλές δυσκολίες. Δύο ερωτήσεις. Μήπως ένα εκατομμύριο υπογραφές είναι πολλές εγώ έχω την, το συνέστημα ότι ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός. Ίσως σε ορισμένα μέρη πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των υπογραφών. Ίσως και αυτό θα το αναφέρω στην έκθεσή μου. Ύστερα, ε, μήπως ο χρόνος είναι λίγος, μήπως πρέπει να τον επιμικίνουμε. Ένα από τα θέματα τα οποία έχω σκεφτεί και ο κύριος Χάφνερ και άλλοι ανέφεραν το θέμα, είναι η εξακρίβωση των υπογραφών. Ε, μου φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν 28 διαφορετικοί τρόποι εξακρίβωσης της ταυτότητας των ατόμων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει, υπάρχει βεβαίως ένα εκλογικό μητρό, αλλά δεν μπορείτε να εξακριβώσετε πολλά πράγματα. Εγώ έχω το συνέστημα ότι, ε, ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ε, ψηφιακό μητρό ε, να δούμε που έχει εισαχθεί. Στην Εστονία έχει εισαχθεί ανεξάρτητα του που βρίσκεται το άτομο. Γιατί να μην γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως θα έχουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια που θα υπερβαίνει, που θα είναι πάνω από την εθνική ηθαγένεια και θα μπορούμε να δούμε αν υπάρχει μια γεραρχία κλπ. Νομίζω ότι πρώτον θα πρέπει να μην είναι υποχρεωτικό αλλά να είναι ε, προαιρετικό αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία ή σε άλλη δραστηριότητα ε, θα πρέπει να κάνει μια απλή αίτηση. Δεν πρέπει, θα πρέπει να είναι ένα απλό έγγραφο ε, να μην περιλαμβάνονται τα πάντα, η ομάδα αίματος και λοιπά αυτό οδήγησε στο, και στην αποτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ταυτότητα. Αυτό είναι θέματα αρχής. Νομίζω ότι κάτι έχει λεχθεί σιωπηρά και ρητά. Η πρωτοβουλία είναι μόνο ένας θεσμός που κινητοποιεί, είναι και κάτι το νομικό και πολιτικό. Πρέπει να είναι τα πάντα θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με όλα αυτά τα κριτήρια. Εάν ένα εκατομμύριο άτομα έχουν ε, λάβει τον κόπο να υπογράψουν και η απόρριψή τους θα δημιουργήσει ένα εκατομμύριο ευρωσκεπτικιστές. Ίσως υπερβάλλω, αλλά πάντως βλέπετε που το πάω. Δημιουργεί απογοήτευση. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί ας πούμε η πρωτοβολία μας έχει απορριφθεί. Και μετά αισθανόμαστε μια απογοήτευση θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα πιο ε, ισχυρό με ακροάσεις ε, για την πρωτοβουλία και ένα θέμα κοινοβουλευτικό είναι σε ποια επιτροπή και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μια ουδιαίτερη ε, επιτροπή ή αναφορών ή αύκο είμαστε οι πιο κατάλληλοι και οι δύο μαζί αλλά όχι απαραίτητα η επιτροπή η οποία είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη διότι θα έχει αντίθετο ίσως συμφέρον για το θέμα. Μ' αρέσει η ιδέα του Συμβουλίου μια φορά το χρόνο ή πιο συχνά θα πρέπει να επιληφθεί το Συμβούλιο του θέματος. Δεν πρέπει να λέει δεν μας αφορά. Ε, πρόκειται για τους πολίτες του Συμβουλίου, για τους πολίτες μας. Θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπε ο συνάδελφος το νομικό κλίμα Ε, ο νόμος επιδέχεται ε, πολλές ερμηνείες. Θα πρέπει το νομικό κλίμα να είναι ευνοϊκό, να διατίθεται ευμενός απέναντι ε, στην ΠΕΠ. Και πάλι τα όσα είπε ο Πατζάκ. Νομίζω ότι ο ρόλος της Επιτροπής και μεταφράζω τα ουγγρικά του στα αγγλικά μου είναι ο πρώτος αξιολογιστής που συνέβαλε ε, στην απογοήτευση που προκάλεσε η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Μπεατρίς Μπετσέρα από την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω την τιμή να είμαι η τελευταία που θα παρέμβει στη συζήτηση αυτή και ίσως έχω το πλεονέκτημα να συνοψίσω όλες αυτές τις ιδέες, τις ιδέες που ακούσαμε σήμερα. Νομίζω ότι ε, ήταν από τις πιο ζωηδές και ζωντανές συζητήσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει. Και πρέπει όλα αυτά να χρησιμεύσουν στον τελικό σκοπό, δηλαδή να επεξεργαστούμε μια έκθεση για την υλοποίηση του κανονισμού για τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών, διότι οι πολίτες, οι συμμετέχουν σε αυτό από την ε, γέννηση της διαδικασίας αυτής. Και θα έχουμε και τις εκθέσεις ε, και των δύο επιτροπών, και ΑΦΚΟ και ΠΕΤΗ. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή ε, θα πρέπει, νομίζω ότι θα είναι, και συγχωρέστε μου την αισιοδοξία, ότι θα είναι αποτελεσματική. Πρέπει να επιλύσουμε ένα, ένα πρόβλημα που υπάρχει, το έχουμε σημειώσει όλοι, και, και μιλούμε για ένα μέσο της βελτίωσης της συμμετοχικότητας των πολιτών, απέναντι σε ένα μέσο που είναι γεμάτο εμπόδια, που λείπουν κίνητρα για τους πολίτες, που δεν καταλήγει σε επιτυχία, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και όλα αυτά <clears throat> δεν μεταφράζονται σε τροποποίηση της πολιτικής ατζέντα σε σχέση με τα αιτήματα που θέτουν οι πολίτες. Αυτό που είναι βέβαια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά συγκεκριμένα μέσα και θα τα προτείνουμε στην έκθεση αυτή και γι' αυτό θεωρώ ότι οι αναφορές πρέπει να είναι στη βάση της υλοποίησης των προτάσεων αυτών στο κέντρο και θα συμφωνήσω με τον κύριο Σεπφλίν ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι σαν ενιαία θηρίδα γιατί στις περισσότερε ε, χώρε έχουμε εκπρο... Ε, εκπροσώπηση της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Αυτές οι θηρίδε θα πρέπει να είναι θεσμικές και ενιαίες, ώστε οι υποδομές που ήδη υφίστανται να χρησιμοποιηθούν, ώστε να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση όλες οι όλοι οι πολίτε των χωρών για το τι μπορούν και το τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να συμμετάσχουν. Θα πρέπει να παρακολουθούμε λοιπόν την προσπάθεια που καταβάλουν οι πολίτες, θα πρέπει να τους συνεπικορούμε νομικά και διαδικαστικά και θα πρέπει να τους προσφέρουμε πρόσβαση με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Και θα πρέπει επίσης να προσφέρουμε κίνητρα και να αυξήσουμε τη διαφάνεια και την ενημέρωση την ενημέρωση ευρύτατα γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζουν οι πολίτες πώς λειτουργούν οι διαδικασίες αυτές και τι συμβαίνει. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και στη συλλογή και στην ε, επικύρωση των υπογραφών. Και εδώ μιλούμε για τους Ευρωπαίους πολίτες και επομένως μιλούμε στην ουσία για την ευρωπαϊκή ταυτότητα Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να λειτουργήσει αν υπάρχει, αν εν υπάρχει ένα τεχνικό εμπόδιο που είναι διαφορετική διαδικασία εξακρίβωση των υπογραφών μεταξύ ε, των χωρών. Αυτό ήταν ένα εμπόδιο που ήταν από τη γέννηση του μέσου της διαδικασίας εκεί και πρέπει να αρθεί. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυόμεθα ισότιμη μεταχείριση σε όλους του πολίτες από όλε τι χώρες και διευκόλυνση της διαδικασία. Τα ψηφιακά μέσα που έχουμε στη θέση μας είναι βέβαια. Είναι βέβαιο ότι τεχνικά μπορούμε να προσφέρουμε ένα πιο εύκολο τεχνικό μέσο ομοιογενές και ισότιμο για όλες τις χώρες, το οποίο θα δίδει τη δυνατότητα μια ενιαία καταγραφής ενό ενιαίου μητρώου τέτοιων πρωτοβουλειών και οποιασδήποτε άλλη πρωτοβουλία και προσπάθεια των πολιτών. Επίση, θα πρέπει οι πολίτε που δεν βρίσκονται στη χώρα του να μπορούν να υποστηρίζουν τέτοιε πρωτοβουλίε. Και θα αναφερθώ επίση απλώ στο θέμα τη ε, πολυγλωσία. Είναι πολύ σημαντικό μαζί με τους εταίρους μας όπως η ΕΟΚΕ να έχουμε μετάφραση των υποβολών και των πρωτοβουλίων αυτών σε όλη τη διαδικασία. Επομένως προκειμένου αυτή η δράση όπως έλεγαν και οι συνάδελφοι από την change.org θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας σε εταίρους και συνεργάτες και όχι μόνο πρέπει να είναι εύκολο και χρήσιμο αυτό που θα κάνει ο πολίτης αλλά θα πρέπει ο πολίτης να ξέρει ότι θα έχει μία τελική σκοπιμότητα. Θα πρέπει λοιπόν η προσδοκία της ε, δυνατότητας αλλαγής των, του νομοθετικού πλαισίου να είναι πραγματική. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ για τη συνεισφορά όλων των σημερινών ε, ομιλητών και, θα, και δεσμεύομαι ότι θα συμμετάσχω σε μια έκθεση που θα διευκολύνει και που θα βελτιώσει αυτή την κατάσταση και που δεν θα είναι ένα κενό ή θεωρητικό γράμμα. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Αν μπορείτε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας. Μάικλ Βαντεμάστ εγώ υπήρξα συντονιστής για μία από αυτές τις πρωτοβουλίες στην Ολλανδία. Σήμερα το πρωί άκουσα πάρα πολλές παρατηρήσεις σχετικά με τα προβλήματα που είχαμε με τη συλλογή των υπογραφών, διάφορα λαθασμένα πράγματα ή ανακριβή που ακούστηκαν. Αλλά θα μπορούσα να μπορώ να πω στους 30.000 ανθρώπους στην Ολλανδία που υπέγραψαν τις ε, αναφορές μας ότι υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί ο ευρωσκεπτικισμός που έχει αναπτυχθεί πλέον. Και νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα από τα παραδείγματα όπου φτάσαμε τουλάχιστον στη δική μας πρωτοβουλία σε απτές νομικές προτάσεις και απερίφθη από τον ίδιο θεσμό που την, που την κατεχώρησε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το εξηγήσουμε τους πολίτες. Ότι οι πολίτες πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν εμπιστοσύνη, πίστη στο σύστημα όταν συμβαίνουν αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούσετε και αισιόδοξα μηνύματα. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, η, η τάση μετά από όλα αυτά που θα ε, παραμείνει είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Ήμουν συνδιοργανωτή σε μια ΠΕΠ. για το βασικό εισόδημα. Τώρα όλοι μας συμβουλεύουν να μην κάνουμε σχετική ΠΕΠ. Να περιμένουμε πρώτα την θετική μεταρρύθμιση τον ΠΕΠ με τις 12 συστάσεις που την ε, υποστηρίζουν όλοι. Και διαβάστε το σχετικό κείμενο που υπάρχει και στο διαδίκτυο. Είναι και ο Κάρθεν στο λόμπι αυτό, από ό,τι φαίνεται. Είμαι και εγώ από την ε, Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών και ε, Πρωτοβουλειών Πολιτών και εκπροσωπώ και ε, μια πρωτοβουλία για την διεθνή δημοκρατία κλπ. Μια ερώτηση. Εμείς έχουμε υποβάλει συστάσεις μετά από μια μελέτη που κάναμε με τις νομικές υπηρεσίες εδώ στις Βρυξέλλες με μια νομική εταιρεία νομικών συμβούλων. Πρέπει να δούμε τον έλεγχο του νομικός παραδεκτού. Θέλαμε να δημιουργήσουμε και έναν ειδικό ε, υπάλληλο για τις ΠΕΠ. Είναι σημαντικό να υπάρχει θεωρούμε γιατί θα εξωτερικεύει αν θέλετε τον έλεγχο του παραδεκτού που είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι περίεργο που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ο τελικός αποδέκτης αλλά και ο φορέας που ε, καθορίζει το παραδεκτό ή μη μιας ΠΕΠ. Αν πούμε ότι, αν πει, αν μια ΠΕΠ στοχεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε πρέπει ο έλεγχος του παραδεκτού να γίνεται από εξωτερικών. και ενδεχομένως να γίνεται ένας διάλογος με τους ενδιαφερομένους. Ε, αυτό ισχύει για τις εταιρείε. Γιατί λοιπόν να μην ισχύει κάτι παρόμοιο με και στην περίπτωση των πολιτών που υποβάλλουν μια ΠΕΠ. Θα μπορούσε να γίνει ε, ένας δομημένος διάλογος με τα άλλα θεσμικά όργανα για τον έλεγχο του παραδεκτού ή ενδεχομένως να υπάρξει από εξωτερικών ο έλεγχος του παραδεκτού. Είμαι Μεζίλ Μπορτελέζα. είμαι ε, μέλος ε, του κόμματος και δεν αναφέραμε σαφώς, ε, δεν έχουμε δει τον ρόλο των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόση εξουσία πρέπει να έχουν πόσες δυνατότητες. Είναι μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει εδώ σχετικά με τον ρόλο που θέλουμε να παίξουν οι πολίτες. Είναι βεβαίως δεν είναι για, για τα τεχνικά θέματα, για το πόσες υπογραφές. Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, διότι δεν νομίζω ότι είναι κάτι που έχει γίνει αρκετά όταν άρχισε να ορισμένοι είπαν α κάνουμε ένα μοντέλο επιχειρηματικό. Μίλησα με ανθρώπους και είπαν ότι θα παρέχουμε τον ΠΕΠ ως υπηρεσία. Και μετά τα εγκατέλειψαν. Μίλησαν με τους πελάτες και τους είπαν μην κάνετε μια πρωτοβουλία που δεν θα επιτύχει. Αυτό συνέβη αρκετά νωρίς. Οι άνθρωποι ε, προσπαθούσαν ε, να βάλουν την ΠΕΠ στο λογισμικό, ε, να μην κάνετε τους ΠΕΠ, τους είπανε κάνετε λόμπι, μιλήστε με τους βουλευτές, μην ασχοληθείτε με την πρωτοβουλία. Αυτό έχει λεχθεί. Ευχαριστώ. Υπάρχει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να λάβει τον λόγο. Όχι. Α, με απογοητεύεται. Είμαι επίσης πολίτης, με ακούτε. Είμαι, ήμουνα σε μια επιτροπή που ήταν για την τορίο ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων και θέλω να απαντήσω στα αυτά που είπε ο κύριος ο προλαλής και οι, οι δύο εισηγητές από την Επιτροπή Πέτη και την Επιτροπή Αυκομαρέση η ιδέα να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες και επίσης η δημιουργία ενός ε, γραφείου εθνικού. Δεν ξέρω βεβαίως αν αυτό θα βοηθήσει πολύ, αλλά νομίζω ότι οι καλύτεροι για να διαδώσουν το μήνυμα είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν υπάρχει έλλειψη γνώσεων, δεν υπάρχει έλλειψη αρμοδιοτήτων για το πώς κανείς να οργανώσει μια πρωτοβουλία. Είναι οι εμπειρογνώμονες ήταν ε, μεταξύ τριών στην Ευρώπη που μπόρεσαν να εγκαταστήσουν λογισμικό ε, και έχει αυτό στην αρμοδιότητα, αλλά δεν επιτύχαμε για άλλους λόγους που αναφέρθηκαν όλοι και περιλαμβάνονται στις ε, δέκα συστάσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Μπέρκ. Μ' αρέσει η δέσμευσή σας να έχετε μια αναθεώρηση ε, του κανονισμού σας. Νομίζω ότι το σημαντικότερο θα ήταν να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις δέκα συστάσεις τροποποιημένες. Αν θέλετε να διαδώσετε το μήνυμα θα πρέπει να σκεφτείτε μερικά μέσα για να υποστηρίξετε τους ίδιους τους πολίτες στο ώστε να διαδώσουν το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι παρούσα από την αρχή του πρωινού, αλλά έχω απλώς μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον αρμόδιο για να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ε, έγιναν πάρα πολλές παρατηρήσεις, συστάσεις σχόλια τα οποία ακούσαμε εδώ και τρεις ώρες πριν από την έγκριση νέου κειμένου η Κομισιό θα παραχωρήσει μια νέα πρωτοβουλία ή θα πρέπει να περιμένουμε με ένα χρόνο όπου δεν θα υπάρχουν αναφορές διότι ε, νέες πρωτοβουλίες, με συγχωρείτε. Διότι αν υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες, ίσως κινδυνεύουν οι πολίτες να απορριφθούν αυτές. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δοκιμάσουμε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εδώ μπορούμε να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κανείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει, όχι. Καλώς. Τώρα περιμένουμε την έκθεση της Επιτροπής η οποία θα λάβει υπόψη τις διαβουλεύσεις, τα σχόλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δούμε αν υπάρξει βελτίωση. Η συνήθις διαδικασία είναι να πούν ότι υπάρχει δυνατότητα ε, τροποποίηση του κανονισμού για να γίνουν οι βελτιώσεις. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν οι ΠΕΠ στο μεσοδιάστημα, δεν θα ήταν κάτι τέτοιο θεμητό αλλά μπορεί να, υπάρξει, να υπάρξουν κάποιοι δισταγμοί από την πλευρά των οργανωτών που θα περιμένουν ίσως μια πιο δεκτική νομοθεσία για αυτούς που θα τους διευκολύνει. Ε, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτό, δεν ξέρουμε. Είναι βέβαια ένα θέμα. Τώρα, οι εισηγητές θέλουν να πούν δύο λόγια και να σχολιάσουν τις κάποιες παρατηρήσεις. Ο Κάρλο Καζίνη. Απλώς να επαναλάβω την απόλυτη βεβαιότητά μου ότι μόνο μια συζήτηση με ψήφο και με την συμμετοχή όλων των βουλευτών και όλων των ε, πολιτικών ομάδων θα μπορέσει να δώσει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν είναι να γίνει με κάποια μεταρρύθμιση, ξαναλέω ότι πρέπει να τροποποιήσουμε τα άρθρα 10 και 11. Και να είναι υποχρεωτική η συζήτηση και η εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοίχω προ τι αναφορέ. Χρειάζεται λοιπόν μια πρόσκληση προς την Κομισιόν που να μην είναι έτσι γενικώ μια πρόσκληση αλλά υπό προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ. Έχουμε άλλα σχόλια, λέει η Πρόεδρος όχι. Συμφωνούμε όλοι μαζί σας. Υποθέτω και είμαι βέβαιη. Θα ήθελα απλώ να πω δύο λόγια Κάποιοι μιλούν δυνατά στα Ιταλικά όπως συνήθως συμβαίνει λέει η Πρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε πράγματι να πούμε όπως είπε κάποιος ότι βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι για τη CCI αλλά πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά για το μέλλον των ECI. Θα έχουμε την ε, δική μας έκθεση, θα έχουμε και την έκθεση της ε, Κομισιόν και είμαι βέβαιος, βέβαιη ότι και η Σεσίλια συμφωνεί ότι να συζητηθεί αυτό στην Λομέλεια και θα το συζητήσουμε οπωσδήποτε και στις επιτροπές μας όταν θα εξετάσουμε την έκθεση. Θα είναι λοιπόν μια ζωντανή διαδικασία σε επόμενους μήνες και πρέπει για να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι εν κενό που εξετάζουμε το μέλλον των ECI. Βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή και στην Ευρώπη και μιλούμε όλοι για το δημοκρατικό έλλειμμα. Μιλούμε όλοι για την ανάγκη του να υπάρξει απόφαση για το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα έχουμε πολλά τέτοια θέματα και το μέλλον. Δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχε νομιμοποιηθεί από τους πολίτες και μιλούμε για μια περιοχή, μια ήπειρο και τις χώρες μας που, έχουν, που βασίζονται στη δημοκρατική παράδοση. Και πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτό το, αυτός ο θεσμός, αυτή η διαδικασία, αυτό το μέσο που είναι ένα μέσο δημοκρατίας να λειτουργήσει καλύτερα και να έχει μέλλον. Αυτό που και η, η έλεγε ε, ισχύει στην παρούσα δύσκολη κατάσταση. Χρειαζόμαστε μια καλή ισορροπία μεταξύ. Χρειαζόμαστε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Απολύτως και ίσως περισσότερο από ποτέ τώρα. Αλλά χρειαζόμαστε και την άλλη πλευρά της συμμετοχικής δημοκρατίας που επικυρώνει τελικά, νομιμοποιεί όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εκ μέρους τουλάχιστον της Δυτικής μου Επιτροπής βεβαίως και θα δώσω το λόγο στην Σεσίλια γιατί μάλλον και εκείνη θα θέλει να πει δύο λόγια για να μου. Ναι, και εγώ όπως και εσύ θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσους συμμετείχαν στη σημαντική αυτή ακρόαση. Λαμβάνομαι υπόψη τα αιτήματά σας, τις αξιώσεις σας, την απογοήτευσή σας, την ανησυχία σας και με μεγάλη σοβαρότητα θα τα δούμε όλα αυτά. Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι εξαιρετικό μέσο που μπορεί να βελτιωθεί και να βελτιώσει και το διάλογο μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα ζητούμενο. Αλλά ακόμα υπάρχει πολύ περιθώριο βελτιώσεων να γίνει πιο φιλικό προς το χρήστη, να είναι πιο εύχριστο. Παράλληλα όμως πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών δεν μπορεί, δεν γίνεται να υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για οτιδήποτε. Ούτε μπορείτε να περιμένετε από το Κοινοβούλιο να δέχεται οτιδήποτε προτείνεται. Υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τα σεβόμεθα. Αυτοί είναι βασικοί κανόνες της κοινοβουλευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ενώ εργαζόμεθα για να γίνει το μέσον αυτό πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς το χρήση. Υπάρχουν δυνατότητες πολλές και πάλι ευχαριστούμε που ήρθατε και μοιραστήκατε τις εμπειρίες και ιδέες σας μαζί μας.